Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται στο φάκελο των Ευρωβουλευτών. Εάν δεν υπάρξει κάποια ε, αίτηση για αλλαγή εγκρίνεται η μερίσια διάταξη χωρίς ε, να τροποποιηθεί. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι για αύριο το απόγευμα έχει ακυρωθεί η συνεδρίαση. Επομένως η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί και το απόγευμα και αύριο το πρωί. Και να σας υπενθυμίσω ότι θα γίνει και μία έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο 7 με 9 στην οποία συνεδρίαση θα γίνει η ψηφοφορία της έκθεσης της συναδέλφου Δελκαστήγιο. Ο κύριος Λάγκεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, μία παρατήρηση να κάνω για την, ε, για διαδικαστικά. Αύριο αλλάζει Έχουμε την προθεσμία για την καταθέση τροπολογιών για την ε, οδηγία για την πρόληψη πλαστικών αποβλήτων. Αύριο λοιπόν η προθεσμία λίγη. Σήμερα η αρμόδια επιτροπή για το περιβάλλον θέλει να αποφασίσει, να ψηφίσει. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια μεγάλη παρατυπία και θα πρέπει η Επιτροπή μας να διαμαρτυρηθεί. Πολύ απλά δεν τηρούνται οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν επειδή η πράσινη εισηγήτρια από τον ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν είναι υποψήφια για τις επόμενες ευρωεκλογέ να μας ε, τρέχει έτσι. Και κατά δεύτερον, κυρία Πρόεδρε, προς μεγάλη μου χαρά χτες ανακοινώθηκε από την Γραμματεία ότι οι τροπολογίε στη δική μας Επιτροπή μέχρι αύριο μπορούν να κατατεθούν μόνο στα αγγλικά. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην γίνονται έτσι σεβαστά τα δικαιώματα των ε, εισηγητών. Αυτό το αποφάσισαν οι σκιώδεις. Είναι δυνατόν να αποφασίζουν οι σκιώδεις εισηγητές σε ποια γλώσσα θα καταθέσουμε τις τροπολογίες μας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, να καταγγείλουμε την απόφαση της Επιτροπής του Περιβάλλοντος και θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη σοβαρά. Ευχαριστούμε κύριε Λάγκεν. Συμφωνώ απολύτως. Η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Επομένως θα στείλουμε αμέσως επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία ετοιμάζουμε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα την κοινοποιήσουμε και ε, στον Πρόεδρο και σε όποιον άλλον πρέπει να ενημερωθεί για την κατάσταση. Ωραία, να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Σήμερα το πρωί έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή Γιάν Σμίτς, ο οποίος θα μας ε, ενημερώσει για την κατάσταση όσον αφορά το πρόγραμμα ε, ορίζοντας 2020, τις εργασίες που κάναμε στη διάρκεια του περασμένου έτους ε, και μετά την παρουσίασή του θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις και να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας. Παρακαλώ κύριε Σμίτς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαρτόρη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια για την κατάσταση της εφαρμογής του Ορίζοντα 2020, διότι όπως αγνωρίζετε έχει ξεκινήσει η πρώτη διαδικασία υποβολής ε, ε, προσφορών ε, το Δεκέμβριο ήδη και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερχόμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας, πώς προχωρούν οι πρώτες υποβολές προτάσεων και πώς λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις σας όλα τα σημεία για τα οποία επιμείνατε. Στη διάρκεια λοιπόν της σύντομης παρουσίασής μου θα αναφερθώ σε κάποια θέματα στα οποία επέμεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας ε, ε, δείξω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής τηρούμε πλέον την διοργανική συμφωνία η οποία επετεύχθη για τον ορίζοντα 2020 και προσπαθούμε να τηρήσουμε όλα όσα έχουν συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ορίζοντας 2020 είχε εξαιρετικά καλή υποδοχή και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτή την κοινή προσπάθεια. Πολλοί από εσά συμμετείχατε στις εκδηλώσεις που είχαμε για την έναρξη του προγράμματος σε κάποιες χώρες. Ε, υπήρχε ο, ο συνάδελφος ο οποίος ήταν παρόν στη Γερμανία και πολλά άλλα, ε, ε πολλές άλλες εκδηλώσεις ε, έγιναν και υπήρξε πολύ καλή υποδοχή και από τους ερευνητές και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εξειδικευμένες οργανώσεις Φαίνεται λοιπόν ότι όλοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα. Και αυτό ε, θεωρώ ότι έχει γίνει χάρη και στην πολύ καλή δουλειά ε, που έχει κάνει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού και έχουν διαμορφώσει το πρόγραμμα αυτό. Είχαμε μια πολύ καλή αύξηση στον προπολογισμό. Ίσως τα 100 δισεκατομμύρια που θα ήθελε το Κοινοβούλιο δεν τα έχουμε καταφέρει μένα, αλλά έχουμε μια σημαντική αύξηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα, διότι η καινοτομία είναι το μόνο τμήμα ενός ε, ε, συρρυκνούμενου προπολογισμού το οποίο αυξάνεται. Και η επιστήμη και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικά και δίνεται και ένα ε, ψυχολογικά πολύ καλό μήνυμα διότι ακόμα και σε ένα συρρυκνούμενο προπολογισμό αυξάνουμε τον προπολογισμό για την έρευνα και την καινοτομία. Θέλουμε να έχουμε ε, περισσότερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και νομίζω ότι με τον ορίζοντα 2020 έχουμε μια πολύ καλή απλούστευση των διαδικασιών και μπορούμε να έχουμε μια καινοτόμα προσέγγιση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να κάνω κυρία Σαρτόρη είναι να διατρέξουν εντάχει τα διάφορα σημεία στα οποία εσείς εδώ στην Επιτροπή σας προσδίδετε ιδιαίτερη σημασία και να σας πω επακριβώ τι κάνουμε αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα στοιχεία. Θα ξεκινήσω με την πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζει ο Κρίστιαν Έλερ, την ε, ε, καινοτομία Fast Track. Ε, στον ορίζοντα 2020 είπαμε ότι αυτό θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, καινοτομία Fast Track και θα γίνει το 2015, το 2016 και εμείς από πλευράς μας δεν περιμέναμε να φτάσουμε στο 2015. Διοργανώθηκε ήδη ένα εργαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου προκειμένου να διαμορφώσουμε λίγο το περιεχόμενο αυτό του ε, πιλωτικού προγράμματο. Η Κρίση Ανέλη συμμετείχε, είχαμε πάνω από 30 ενδιαφερομένους και έχουμε δεσμευθεί να έχουμε αποτελέσματα, να δαπανίσουμε αυτά τα 100 εκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί για αυτό το πρόγραμμα μέχρι το 2020 και συνολικά 200 ε, εκατομμύρια για αυτή την πιλωτική πρωτοβουλία. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν, έχουν ε, ληφθεί οι πρώτες πρωτοβουλίες για να δοθεί μορφή σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε και ιδιαίτερη υπομονή, επιμονή σε συγκεκριμένα μέσα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περισσότερο προπολογισμό, περισσότερη προσοχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο Φιλίπ Λάμπερτ έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία που να ασχολείται με τα θέματα αυτά, δεν θα πρέπει να τα κατανέμεται σε διάφορες υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση, αλλά τίναμε βίκονους και δημιουργήσαμε μια ειδική υπηρεσία που θα ασχολείται με το θέμα αυτό. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως ε, στο θέμα αυτό το οποίο ε, ενδιαφέρει τον Φίλιπ Λάμπερς, να υπάρχει ειδική υπηρεσία που να ασχολείται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πρώτες προσκλήσεις ε, για τους διαγωνισμούς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 560 εκατομμύρια έχουν ήδη διατεθεί σε μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στις προκλήσεις του 2014 και 2015. Δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη προτεραιότητα στα θέματα αυτά και θέλουμε να είναι πλήρως επιτυχημένα και να σεβαστεί πλήρως και όλα όσα έχει υποδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον προϋπολογισμό δηλαδή που θέλουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από ό,τι θυμάμαι στις συζητήσεις εδώ, το Κοινοβούλιο επέμενε πάρα πολύ για τα θέματα ενέργειας και η ενέργεια ε, θεώρησε ότι θα πρέπει να την χάνει ιδιαίτερης προσοχής. Η κυρία Μαντουρέλ ε, και ο, ο κύριος Ζαν ε, Πιεροντή επέμεναν για τα θέματα αυτά, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει έρευνα για την ενέργεια. Και γι' αυτό ακριβώς στις πρώτες προσκλήσεις διαγωνισμών που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο ε, το έχουμε θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και σεβόμαστε και ε, το 85% με 15% του προϋπολογισμού. Αυτές είναι οι υποδείξεις που είχατε δώσει εσείς για τα μη ορυκτά και ορυκτά καύσιμα και εμείς λοιπόν στις πρώτες προσκλήσεις ε, έχουμε σεβαστεί αυτό το αίτημα και δημιουργούμε μία σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικό τομέα για τα ε, ορυκτά καύσιμα και το υδρογόνο και φυσικά αυτό θα είναι και σημαντική συνεισφορά και λαμβάνουμε υπόψη και τους στόχους του 15% που έχετε θέσει και έχουμε τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις και τα έχουμε προβλέψει αυτά στα πλαίσια των πρώτων προσκλήσεων. Έγινε επίσης μια μακρά συζήτηση για τη διεύρυνση τη συμμετοχή εδώ στην Επιτροπή σας και ένας από τους πρώτους ε, που συνεισέφεραν ήταν ε, ο κύριος Ρόιλ. Και αυτό λοιπόν το έχουμε πλέον μεταφράσει σε μια προτεραιότητα μέσω αδελφοποίησης, μέσω ενίσχυσης εθνικών σημείων επαφής. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σε αυτή την πτυχή της διεύρυνσης και την άνοιξη Στη Βαρσοβία θα υπάρχει και μία συνεδρίαση αφιερωμένη σε αυτό το σκοπό για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ε, περισσότερη διεύρυνση για να μπορέσουμε να ε, πληρώσουμε αυτό το χάσμα της γνώσης που υπάρχει στην Ευρώπη. Από αυτή την πλευρά λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό το θέμα αποτελεί προτεραιότητα και κυρίως στον τομέα της αδελφοποίησης ε, μεταξύ ε, μεγάλων ε, ερευνητικών ιδρυμάτων στις, σε διάφορες περιοχές Ευρώπης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη κάποια ε, θετικά στοιχεία και αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε και τη δέουσα σημασία. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι ο κύριος Φανίστερο επέμενε ιδιαίτερα ε, για το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή και προσέχουμε και εμείς αυτό το σημείο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιστήμη με και για την κοινωνία. Είναι ένα στοιχείο επίσης που εσείς στην Επιτροπή σας ε, το ε, θεωρήσετε ιδιαίτερα σημαντικό. Ζητήσετε και σχετική γραμμή προπολογισμού. Έχουμε ξεκινήσει εκεί και κάποιες προσκλήσεις το Δεκέμβριο όπως σας είπα και πάλι το θεωρούμε προτεραιότητα. Έχουμε ήδη τέσσερις προσκλήσεις στον τομέα αυτό και επομένως και από αυτή τη σκοπιά έχουμε τηρήσει τις υποχρεώσεις μας διότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι ε, η επιστήμη και η εκπαίδευση και η καριέρα σε επιστημονικούς τομές είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κυρία Πιλάρ Δελκαστήγιο και πολλοί άλλοι εδώ στην Επιτροπή αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά και εμείς από πλευράς μας ε, είπαμε ότι αν δεν υπάρχουν και κοινωνικές επιστήμες οι οποίες θα συμπεριληφθούν πλέον στην έρευνα διαδικασία δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα ε, απόλυτα. Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα στις πρώτες προσκλήσεις ε, ε, για διαγωνισμούς όπου συμπεριλαμβάνονται κοινωνικά θέματα στον τομέα της υγείας, στον τομέα των μεταφορών. Και εγώ θα ήθελα ίσως να πάω και ένα βήμα περαιτέρω στο δεύτερο γύρω προσκλήσεων ε, προσφορών. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να ε, συμπεριλαμβάνουμε το θέμα, αλλά έχουν να γίνουν και άλλα, ε, και άλλα προς αυτό το σκοπό. Τα θέματα φύλου. Πολλοί από εσά θεωρήσατε ότι θα πρέπει να επισημάνουμε και τη διάσταση του φίλου και ε, θέλετε να λάβουμε υπόψη ε, τη διάσταση του φίλου και πρέπει να σας πω ότι οι συμβουλευτικές ομάδες που συστήνονται δεν έχουν στόχο το 40% αλλά το 50% και έχουμε καταφέρει στο 50% των μελών των συμβουλευτικών ομάδων να έχουμε γυναίκες ερευνήτριες ε, από το δημόσιο και από το ιδιωτικό τομέα. Και ήταν ενδιαφέρον αυτό, διότι αρχικά εσωτερικώς είπαμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά μετά είπαμε ας μην δοκιμάσουμε το 40%, δοκιμάσουμε 50% και τα καταφέραμε και χωρίς πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι καλή ένδειξη και δείχνει και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, καταφέρει αυτά τα οποία τη ζητάτε. Ε, και αυτό θα σας το αποδεικνύω κάθε φορά όποτε μου επιτρέπετε να σας δείξω ότι όντως ε, ακούσαμε τι έχετε να μας πείτε και θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Θεωρούμε ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε θέματα φύλου και διευκρινίζουμε σαφώς ότι σε κάθε πρόσκληση που λαμβάνουμε οι συμμετέχοντες και οι ετούντες θα πρέπει να μας υποδείξουν πώς λαμβάνουν υπόψη και τα θέματα του φύλου. Αυτό είναι καινοτομία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική καινοτομία να δημιουργηθεί μια νοοτροπία ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτά τα θέματα. Η κυρία Μαντουρέλ και η κυρία Καρβάγιο ζήτησαν να υπάρχει και ε, επιστημονικό πάνελ για την υγεία. Ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Έγινε μια συνεδρίαση. Ε, θα γίνει και άλλη συνεδρίαση μέχρι το τέλος του μηνός. Γίνεται κάποια πρόοδος, αλλά είναι πιο περίπλοκο από ό,τι περιμέναμε. Θα τα καταφέρουμε όμως. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Η απλούστευση. Το είχαμε αναφέρει αυτό στον ορίζοντα, στον το 2020. Νομίζω ότι όλοι εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή έχετε απευθύνει έντονη έκκληση για την απλοποίηση αυτή. Θα πρέπει να βγούμε από την ε, μικροδιαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση ε, με σωστή βάση για ένα ενιαίο πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε γρηγορότερες επιδοτήσεις σε 8 μήνες. Η κυρία Καρβάλιο νομίζω έκανε και κατήρθησε ένα κατάλογο με 58 ε, σημεία και λοιπόν ε, τα λάβαμε όλα υπόψη και νομίζω ότι τα εκτελέσαμε όλα αυτά και νομίζω ότι ε, σε θέματα απλοποίησης τα πήγαμε καλά. Φυσικά ο διάολος κλείβεται στις λεπτομέρειες και παρακολουθούμε στενά το θέμα αυτό προκειμένου να είναι όντως η πρόσβαση στα προγράμματα πιο εύκολη, να σεβόμαστε τα χρονοδιαγράμματα για τις ε, επιδοτήσεις και προκειμένου να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες για την απλοποίηση. Άρα, σε όλα αυτά όντως ακολουθούμε τους στόχους μας και το χρονοδιάγραμμα. Αυτά λοιπόν συνοπτικά κύριε Σαρτόρη. Δεν θέλω να σας απασχολήσω και να μακρηγορήσω πιο πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι από πλευρά της Επιτροπής σεβόμαστε απόλυτα αυτά που συμφωνήσαμε και θα έπρεπε σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω ασφαλώς όχι μόνο τα διάφορα θέματα τα οποία ε, αναφέραμε αλλά και μια εμβληματική πρωτοβουλία από, το, ε, από την Επιτροπή, από, την, ε, το Συμβούλιο αυτή, αυτό έρευνας και κοιτώ και προς την πλευρά της κυρίας Αγγέλικα Νίμπλερ η οποία έχει προωθήσει αυτό το θέμα και το έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και πλέον ε, μιλάμε για ένα σχέδιο με 15 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πρικοδότηση. Νομίζω λοιπόν ότι ακολουθούμε αυτά που μας έδωσε ως κατεύθυνση στο Κοινοβούλιο. Πολλά μπορώ να αναφέρω ακόμα για να σας καταδείξω ότι πραγματικά σεβόμαστε την πολιτική συμφωνία. Από δικής μας πλευράς θέλαμε να έρθουμε και να σας παρουσιάσουμε το τι έχουμε κάνει και ότι σεβόμαστε απόλυτα τη θεσμική συμφωνία επί της οποίας έχετε συμφωνήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Διευθυντή. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Καταρχάς ο κύριος Βανίστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις από δική μου πλευράς ε, με όλες τις πρωτοβουλίες, με όλες τις φιλοδοξίες που έχουμε. Τι γίνεται με τις πληρωμές για τη τρέχουσα περίοδο του προγράμματος πλαίσιου. Στη μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχουν καινούργια κονδύλια τι γίνεται όμως με τα leftovers, με τα χρήματα που έχουν μείνει από το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές προς πανεπιστήμια, γιατί θέλω επακριβείς πληροφορίες. Αυτό απασχολεί, ξέρετε, πολύ τον επιστημονικό κλάδο. Μία άλλη ερώτηση. Αυτό που λέτε για την υπηρεσία για τις μικρομεσίες επιχειρήσεις, να προσέξουμε ή να μην διοργανώσουμε καινούργια πράγματα τα οποία ενδεχομένω να μην αποδώσουν. Πείτε μας, εγώ θα ήθελα σε επίπεδο κρατούς μέλους να οργανώνονται αυτά πάρα πολύ καλά. Πείτε μου λοιπόν, δώστε μου πιο πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό. Τι γίνεται στα εθνικά κρατημέλη, στις πρωτεύουσες, αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ίσως να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Τελευταία παρατηρήση τώρα σε ό,τι αφορά την διεύρυνση της συνεργασίας που αναφέρατε. Η συνεργασία που υπάρχει και υφίσταται μεταξύ των προγραμμάτων, μεταξύ των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης μπορεί να επεκταθεί. Τα εθνικά προγράμματα υποβάλλονται, συμφωνούν τα κρατη σε μια εταιρική σχέση σε ό,τι αφορά τέτοια περιφερειακά προγράμματα. Πείτε μας. Γιατί έρχεστε και πριν από τις ευρωεκλογέ εδώ, σε μια ακρόαση σε ό,τι αφορά τέτοια ζητήματα. Πείτε μας λοιπόν πώς θεωρείτε, πώς αξιολογείτε την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών. Υπάρχει κάποια, συνέχιση, σε, κάποια συνέχεια σε ό,τι αφορά την πρακτική τους εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά και την ακρόαση που θα διοργανώσουμε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο το Μάρτιο σχετικά. Ευχαριστώ, κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Σμίτς ε, για την ε, παρουσία του. Είναι πολύ σημαντική, ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντική και η έρευνα και η ανάπτυξη. Καταρχάς λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της υγείας και τη σημασία που έχουμε προσδώσει στο θέμα αυτό. και για τη μείωση των ε, δαπανών ε, για τα φάρμακα, που ορισμένες φορές ε, είναι δυσβάσταχτα. Η έρευνα λοιπόν για μεθόδους ελέγχου των φαρμάκων, εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου των φαρμάκων, ώστε να μπορέσει να μειωθεί και η τιμή τους. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και την πτυχή των ανθρωπιστικών σπουδών. Να επισημάνω δηλαδή το γεγονός ότι προκειμένου να είναι βιώσιμες οι αλλαγές οι οποίες μας περιμένουν, θα πρέπει να ε, μπορούμε να έχουμε και άλλα αγαθά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συνύπαρξή μας. Και είναι το νήμα το οποίο θα μας επιτρέψει γύρω από την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κοινού αγαθού να αναπτύξουμε και κάποια άλλα αγαθά, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά με τα υλικά αγαθά. Αυτή λοιπόν είναι μια ακόμα πτυχή την οποία θα ήθελα να τονίσω, διότι πραγματικά με εκπλήσει η αλλαγή του κλίματος και οι ζημίες που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ της έρευνας για την ενέργεια και της έρευνας για την ε, ε, προστασία του ε, περιβάλλοντος και των εδαφών, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τέλος, ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω διότι άκουσα ότι υπάρχει μια κάποια δυσκολία για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες της JTIs, διότι υπάρχει πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτές τις δραστηριότητες που έχουν ε, βιομηχανικό χαρακτήρα να τις ε, συγκεράσουμε με τα χρονοδιαγράμματα του ορίζοντα 2020 και επομένως θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ ευχάριστο ότι έχουμε εδώ πέρα αυτή την παρουσίαση εδώ στην Ήτρα γιατί είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα είμαστε τα επόμενα χρόνια. Συμφωνώ ότι για την έρευνα, για την ανάπτυξη κάνουμε μετά πρόοδο αλλά να κάτσουμε να ζυγίσουμε πόσα χρήματα έχουμε και τι ανάγκη υπάρχει. Άρα είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους και πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ε, πολιτούς πλαισίου. Γιατί για το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σαφές ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους γιατί για μας ε, αυτού του είδους η καινοτομία fast track είναι φάρμακο κατά της κρίσης. Άρα θα πρέπει εδώ και τώρα να ενεργήσουμε. Επίσης έχει συζητηθεί το γιατί αποφάσισαν ότι αποφάσισαν για τη χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Όμως σας ερωτώ πώς να τον εξασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη να μην παρετηθούν από τους πόρους τους σχετιζόμενους με την έρευνα τα δικά τους χρήματα και να στηρίζονται μόνο στους πόρους από Βρυξέλλες. Θα πρέπει μέρες να εμπλακούν περισσότερο τα κρατημέλη και να βάλουν και αυτά τον βολό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Άλλο. Σας ερωτώ πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε παρά το, ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων να, να μείνουμε πιστοί στο, στις αρχικές μας ιδέες, στις βασικές αρχές αυτές που αποφασίστηκαν στην αρχή. Συγχαρητήρια πάντως γιατί μέχρι τώρα τα έχει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τη διαχείριση των πραγμάτων, των πόρων. Νομίζω ότι πρόκειται για μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο έχετε κάνει. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσία του και επίσης ε, για το γεγονός ότι αυτή η συνεργασία και αυτός ο διάλογος με την Επιτροπή μας ε, ήταν ε, ε, πάρα πολύ σημαντικός. Εκτίμησα ιδιαίτερα και την ταχύτητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα. Όχι μόνο τα όσα λέει δηλαδή το κείμενο, αλλά και την οπτική του και τις ε, προτεραιότητες που είχε υποδείξει η, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή μας και που σέβεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις, διότι το βασικό όραμα, τι αρχές μας κλπ. σας τα έχουμε πει και εσείς σε κάποιο βαθμό τα εφαρμόζετε με κάποια συνέπεια. Πολύ συγκεκριμένες λοιπόν ερωτήσεις. Μία παρατήρηση και σία αν θέλετε, πρόταση. Καταρχάς, προσοχή να μην κάνετε πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό και μην χαθεί η αξία της ε, επιρροής που θα μπορούν να έχει ορίζοντας 2020. Μόλις είπε και η κυρία Χέρτσοκ ότι ορίζοντας 2020 είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν τους χαλεπούς καιρούς της κρίσης. Προσέξτε λοιπόν μην τα κατακαιρματίσουμε πολύ όλα αυτά και χάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και δεν έχουν καμία σχέση με τη σημαντική επιρροή που θα μπορούσε να έχει στον παραγωγικό κόσμο και στην κοινωνία ορίζοντας 2020. Οι ερωτήσεις μου είναι συγκεκριμένες. Πώς μπορούμε να ενημερώσουμε. Κάποιος συνάδελφος έλεγε, μας ρωτάει ο ακαδημαϊκός κόσμος. Εμείς δεσμευτήκαμε, προσπαθήσαμε να γνωστοποιήσουμε τον ορίζοντα 2020, κάναμε και μια δουλειά η οποία δεν μας αναλογεί εμάς. Δεν ξέρω στην Ιταλία εσείς που κάνατε αυτές τις εκδηλώσεις, παρουσίασε αλλά έχω την εντύπωση ότι στη χώρα μου τουλάχιστον υπάρχει μια δυσπιστία, δεν συμμετείχαμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ως χώρα και τώρα ίσως ε, ξεκινά μια νέα διαδικασία, αλλά θα πρέπει να είμαστε και στο ύψος των πληροφοριών που δώσαμε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξή. Πώς οργανώνεστε, διότι όταν μας ρωτάνε πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε κάποιους προσανατολισμούς. Πέστε μας λοιπόν πώς τα οργανώνει η Γενική σας Διεύθυνση τα θέματα του ορίζοντα 2020 για να ξέρουμε πού να τους πούμε να απευθυνθούν, πού να γράψουν, πού να ζητήσουν πληροφορίες. Αυτή λοιπόν η πρώτη ερώτησή μου. Πώς οργανώνεστε για την εφαρμογή όλων των ε, προγραμμάτων. Και αυτή τη στιγμή γίνει η υποβολή των προτάσεων. Πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει την επιλογή. Ε, θα τα δώσετε κάπου εξωτερικά. Για μας είναι λίγο θολά αυτά και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι ένας ευρωβουλευτής δεν ξέρει τι του γίνεται. Και τέλος, ε, τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω, τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά όσο περισσότερες πληροφορίες μας δώστε για τη διαδικασία, τι γίνεται με τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ε, όλα αυτά τα στοιχεία, τόσο πολύ περισσότερο μας μπορέσετε να μας βοηθήσετε να συνεργαστούμε, γιατί ενδιαφέρονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια και θα πρέπει να υπάρχει επίσης όρης αντιμετώπιση. Η κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς κύριε Γενική Διευθυντά καταρχάς ε, για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας για να μας ενημερώσετε για την ε, εξέλιξη του προγράμματος Horizon 2020. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η αρχή και μπορούμε λοιπόν να πάμε και στις εκλογικές μας περιφέρειες να είμαστε έτοιμοι για τις ευρωεκλογέ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα. Έχουν γίνει λοιπόν οι πρώτοι διαγωνισμοί. Είναι πολύ καλές αυτές οι ειδήσει, θεωρώ και μπορούμε έτσι με ευκολία να τις διαβιβάσουμε. Δύο ερωτήσεις να κάνω συγκεκριμένα. Η πρώτη. Να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Τόγια, η συνάδελφος Τόγια. Από διοργανωτικής άποψης, ε, πώς ε, έχετε αλλάξει ε, τα πράγματα στη γενική σας διεύθυνση. Πώς έχει αλλάξει η συγκεκριμένη διαχείριση, η συγκεκριμένη εξέλιξη και εκτέλεση των προγραμμάτων έχει ανατεθεί στις υπηρεσίες όχι μόνο για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, γιατί για αυτές ε, είπατε ότι υπάρχει μια ειδική υπηρεσία πλέον, αλλά και η εφαρμογή, η εκτέλεση των άλλων προγραμμάτων γίνεται μέσω εξωτερικών υπηρεσιών. Τι κρατάτε εσείς ε, στο ιστορικό της υπηρεσίας σας και τι έχετε αναθέσει εξωτερικά. Και ήθελα να ρωτήσω, όπως και συνάδελφο συνάδελφος Τόγια, σε ποιον απευθύνονται συγκεκριμένα τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές, το γνωρίζει αυτό η επιστημονική κοινότητα, σε ποιον δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθεί. Αυτή η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση ρώτησα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματο Εδώ στο Κοινοβούλιο έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την, μετά την, ε, το σκάνδαλο με την ε, NSA. Έχουμε και συλλέγουμε τα σχετικά στοιχεία. Ελπίζουμε να τα έχουμε ολοκληρώσει αυτά αυτή την έρευνα πριν το τέλος της θετίας. Έχουμε το θέμα της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς, το Ευρωπαϊκό Νέφος, το Cloud. και έχει διατεθεί μια, ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο κονδύλι σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά αυτά προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω ε, τι έχει ξεκινήσει ως δραστηριότητα, ως ενέργεια, προκειμένου σε αντίβαρο και προς τη ΣΥΠΑ να κοιτάξουμε την ανεξαρτησία μας σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Έχουν γίνει συγκεκριμένοι διαγωνισμοί. Να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος ε, στις περιφέρειες ε, ρωτάει τι κάνουμε, τι κάνουμε, συγκεκριμένα, τι φτιάχνουμε για την ασφάλεια, για τον κόσμο, για τα δεδομένα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ, ο συνάδελφος Τζόνσον. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σμίτ και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους σας για τα όσα μας είπατε και για την συνεργασία, για τις προτεραιότητες για το Horizon 2020. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για αυτή σας την έκθεση και τη συζήτηση για τις πρόπτικες που κάποιοι θεωρούσαν ότι αποκλείεται να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την ισότητα των φίλων για το 50% Δεν μπορούμε παρά να είμαστε επομένω αισιόδοξοι για το 2020. Έχω κάποιε ερωτήσει, όχι γιατί θέλω να επικρίνω αυτά τα οποία κάνετε, απλώ γιατί θέλω να πετύχουμε ακόμη περισσότερο πρώτα-πρώτα όσον αφορά τι ΜΜΕ. Τι γίνεται με το Eurostar και τις ΜΜΕ. Ε, Είναι το ε, ένα πρόγραμμα να συνδυαστεί με το άλλο. Κάτι άλλο το οποίο είπε ο κ. Φανίτσελ Όσον αφορά τη σχέση ιδιωτικών ταμείων και το ορίζον 2020. Τα κράτη-μέλη δίνεται υψηλότερη προτεραιότητα στα, στις αντισταθμίσεις αποζημιώσεις των διορθωτικών ταμείων. Γιατί κατάθεσαν δυσκολία πολλές εταιρείες. Και δεν προσέχουν τόσο πολύ αυτό το οποίο θέλουν εμείς, δηλαδή την έρευνα και την καινοτομία. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πώς έχει η κατάσταση. Ναι, σύμφωνα με αυτό που λέτε. Γιατί βέβαια αυτό απόκειται στα κράτη-μέλη, αλλά και εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε κάποια δραστηριότητα ως κοινοβούλιο. Επίσης, άλλη ερώτηση. Τι είναι με τον ιδιωτικό τομέα, τι είναι με τις εταιρείε. Είναι πάρα πολύ δραστήριες. Υπάρχει συγχρηματοδότηση όσον αφορά την έρευνα και την κοινοτομία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε και σχέση με αυτό. συνεχίζει να ισχύει αυτή η έντονη δραστηριότητα και η συγχρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό σα λέω τρέφω αισιοδοξία για το μέλλον. Επίση, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, είχαμε πει για την διεύρυνση. Γιατί ε, από πλευρά Σουηδία και άλλων χωρών ξέρουμε ότι η καινοτομία ε, έχει να κάνει με κάποια δεσμικό οργάνωση χώρε μα, αλλά μιλούμε για έρευνα, ε, καινοτομία και δραστηριότητα στην αγορά. Άρα θα υπάρξει διεύρυνση όσον αφορά αυτού του είδους την ε, έρευνα ε, την καινοτόμα και ώστε να υπάρχουν προοπτικές θετικές για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε ακούσει τους μισούς ομιλητές. Κλείνει ο κατάλογος. Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Σμίτ για να δώσει να πρώτο γύρο απαντήσεων για να είναι και πιο απλά τα πράγματα και μετά να ακούσουμε τις υπόλοιπους. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, να τα πούμε σε δύο γύρους. Πρώτο πρώτα μας είπε για τις επιστώσεις πληρωμών ο κύριος Φανίστελρο. Η κατάσταση όντως είναι ενισχυτική διότι θα ξέρετε καλά και η κυρία Χέρτσοκ και ο κύριος Οντή τα είπανε ότι συνεχώς περικόπτει πιστώσεις πληρωμών το Συμβούλιο. και υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικέ πιστώσεις βέβαια με την ολοκλήρωση του 7ου προγράμματος πλαίσιο. 1,1 δις υπολογίσαμε ότι θα μας λείπουν όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Αυτό σημαίνει τεράστια προβλήματα. Χαίρομαι που το είπατε. Ελπίζω και η δική σας επιτροπή και άλλες επιτροπές να προσέξουν το τι θα γίνει. Γιατί είναι σαν να χρησιμοποιούμε τώρα πιστοτική κάρτα. Αναβάλουμε και αναβάλουμε. Αλλά τελικά θα πρέπει να πληρώσουμε. Όλε αυτέ τις περικοπέ του Συμβουλίου θα είναι μεγάλο πρόβλημα σε λίγα χρόνια. Γιατί με μία ΜΜΕ τώρα. Όντω εμεί χρησιμοποιούμε την υπάρχουσα υπηρεσία για αυτό το σκοπό Έχουμε άμεση διαχείριση, δεν συνεργαζόμαστε επομένως με τις εθνικές ε, υπηρεσίες και έτσι επομένως έχουμε υψηλή ποιότητα στη διαχείριση. Τώρα όσον αφορά την ε, διεύθυνση δραστηριότητα σε σχέση με τα διευθυντικά ταμεία και το Horizon 2020 έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε φτιάξει αυτόν τον, ε, τον πάρα πολύ οδηγό για το τι ανάγκες υπάρχουν αλλά τελικά αυτό το οποίο χρειάζεται να διαπιστωθεί είναι ότι τώρα έχουμε 60 με 70 δις από τα διευθυντικά ταμεία. Αυτά έχουν δεσμευτεί για την ε, καινοτομία και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ ε, στενά με τους που και η Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και θα πρέπει επίσης να προσέξουν θα είναι και με τα εθνικά προγράμματα. Έχουμε τα πρώτα σχέδια συμφωνίες σχέσεων, όπως με την Πολωνία, και θα πρέπει τώρα να δούμε το πώς θα καταφέρουμε να έχουμε αρκετέ δραστηριότητε που να καλύπτονται από αυτές τις συμφωνίες θετικής σχέσης. Επομένως, στενή συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση. Ο κύριος Πρόντι Αναφέρει και στα θέματα της υγείας και στο ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, μειώσεις όσον αφορά τις τιμές των φαρμάκων. Έχουμε προτείνει αυτή την εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό το λόγο. IMI. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει για τι ανθρωπιστικέ επιστήμε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται πάντα τα πνευματικά προγράμματα. Όμω η συμβολή είναι πάρα πολύ σημαντική, ούτω ώστε να γνωρίσουμε τι προκλήσει που έχει το συγκοινωνία. Κυρία Χέρτσοκ, αναφερθήκατε σε κάτι που είναι και για μένα εφιάλτη. Οι περικοπές για το για το Ίζον 2020 Έχουμε τις περικοπές, όπως εκείνη την περικοπή, 600 εκατομμύρια φορούν την Ισπανία. Το έχω συζητήσει με τον καθηγητή Μπουργκινιό, ο οποίος ευτυχώς είναι εδώ, από πλευράς Ευρωπαϊκού Χώρου ε, Έρευνας. Και έχουμε τόσο πολλές προτάσεις που κινδυνεύουμε να καταρρεύσει το οικοδόμημα. θα πρέπει και τα κρατημέλη όντως σε περιφερειακό επίπεδο και εθνικό επίπεδο να πληρώσουν, να δοπανίσουν. Εμείς πάντα συνεχίζουμε με την δέσμευση αυτού του περίφημου 3%. 3% του ΕΠ πρέπει να δοπανίσουν τα κρατημέλη σε σχέση με την καινοτομία για το Horizon 2020. Υπάρχει και ένα έγγραφο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις θερινές διακοπές. Θα προέρχεται από τους επιτρόπους Queen και Ρεν. Οικονομική πολιτική, ευρωπαϊκό εξάμεινο, ασχολούνται οι επίτροποι με αυτό εντατικά και έτσι να δούμε τι πολιτική θα ασκηθεί, για την έρευνα και κοινοτομία. Οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κυρία Τόγια. Για τον αντίκτυπο του ορίζοντα 2020. Ναι. Θα πρέπει να έχουμε από τα αποτελέσματα να συνεργαστούμε επιτυχώς με τη βιομηχανία Είναι περίπλοκα τα πράγματα, υπάρχει γραφειοκρατία. Θα πρέπει να τονώσουμε αυτή τη συνεργασία με την βιομηχανία. Με το Horizon 2020 θα ανακτήσουμε την τυχόν απολευθήσα. εμπιστοσύνη. Συνεργασία και με τις ΜΜΕ. Θεωρούν ότι το Horizon 2020 είναι αυτό που περιμένανε. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια. Να ξέρει ο κόσμος σε τι συμμετέχει με το website, με φυλάδια, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς επιλέγονται οι μπειρογνώμονες, φερρυπίν, διαφάνεια να υπάρχει. Και όποιοι υποβάλλουν αιτήσει να το έχουν αυτό υπόψη. Ό,τι και να πω είναι λίγο όσον αφορά την συμμετοχή των εθνικών σημείων επαφής. Αυτή είναι η πρέσβευτες για το ορίζον 2020. Αυτοί θα διαχειριστούν όσους προβάλλουν αιτήσεις στο μέλλον. Τα προγράμματα κλπ. Κύριε Νίβλερ, μας είπατε δύο λόγια για τον οργανισμό. Έχουμε δύο οργανισμούς μέχρι τώρα. Και έχουμε και τον Ευρωπαϊκό χώρο της ε, έρευνας. Αποδίδουμε. Έργο εξαιρετικό. Αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους. Αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ αποτελεσματικές και δεν θέλουμε να συγκροτήσουμε καινούργιες. Θα στηρίξουμε τις υπάρχουσες. Αυτό το αξιόλογο έργο που έχουν επιτελέσει να συνεχιστεί. Επίσης, έχουμε 5% λιγότερο προσωπικό, αλλά έχουμε 20 δις παραπάνω ως προοικοδότηση από τα 30 ανέβηκαμε στα 50 και άρα θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά που μας εμπιστεύονται για όλες αυτές τις αιτήσει τώρα όσον αφορά εγώ θέμα της Ε, υπάρχει αυτή η πρόκληση αφορά την κοινωνία μας, αφορά την ασφάλεια και προβλέπονται κάποιες ε, πρωτοβουλίες τόσο ώστε να, να δούμε τι θα γίνει με την κυβερνοασφάλεια, συνεργασία με την Europol. Οπότε μπορώ να σας ενημερώσω πιο συγκεκριμένα αν θέλετε. Επίσης, ε, όταν, όταν θέλουμε να κάνουμε την πρόσκληση υπο, υποβολής προσφορών, έχουμε πολλά κρατημέλη που μας ε, μπλοκάρουν. Κύριε Γιώχανσεν, μας είπατε για την ισότητα των φίλων Χαίρομαι και εγώ, οπότε για το 40 πήγαμε στο 50%. Άρα εκεί μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα για τις ΜΜΕ μεταξύ Eurostars και του νομοθετήματος για τις ΜΜΕ θα υπάρξει ε, εκεί συμπληρωματικότητα και συμβατότητα. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο σε σχέση με τα ιδιωτικά ταμεία τώρα όσον αφορά την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα όπως προανέφερα ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει συμμετάσχει τόσο όσο θέλουμε σε προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο. Γιατί υπάρχει τρομερή γραφειοκρατία επίσης, γιατί το πρόγραμμα δεν επέτρεπε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, αλλά τώρα καλύπτουμε και την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία. Να, επομένως, το κίνητρο για τη βιομηχανία. Τώρα έχουν κίνητρο να μπουν στο παιχνίδι. Άρα πολλά και το μέλλον και για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και για τις μικρότερες. Χρειάζεται συμμετοχή αυτός ο κλάδος οικονομίας, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο στόχος του προγράμματος πλαισίου είναι να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, το λέει η συνθήκη. Άρα θα πρέπει να εμπλακεί η βιομηχανία. Ωραία. Να περάσουμε στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Έχουμε οχτώ ομιλητές, δύο λεπτά ο καθένα, ο κύριο Βαλέσκη καταρχά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικά και Διευθυντά, καταρχάς να σας πω ότι είχα μήνυμα από το Κοινοβούλιο μου στην Πολωνία δεν είναι ικανοποιημένοι, δεν μπορούν να δεχτούν αυτούς τους τόσο ωραίους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020. Η ανησυχία τους είναι ότι οι ανεπτυγμένες χώρες αναπτύχθηκαν χωρίς να τηρούν όλους αυτούς τους περιορισμούς και εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίσουμε και ζητούν κάτι το οποίο να είναι πιο ρεαλιστικό, να μην είναι απλώς ευσεβής πόθη και να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Ε, να μην πετάμε στα σύννεφα, να μην είμαστε ουτοπιστές και... Ε, φαντάζομαι ότι θα λάβετε και σχετικά στοιχεία αν δεν τα έχετε λάβει ήδη. Επίσης να σας πω ότι εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα ότι έχουμε αυτό τον ορίζοντα, μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Η επιστήμη είναι δύσκολη γυναίκα και χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί, να την ε, δαμάσουμε και ε, καλό είναι που έχουμε ορίζοντα. Και επίσης αυτή η έμφαση που δίνεται στην έρευνα η οποία θα είναι προσανατολισμένη και στη βιομηχανία. Αυτό είναι και καλό και κακό. Η βασική έρευνα η, ε, είναι και πάλι δύσκολη και επομένω δεν ξέρουμε ποιος, πότε, πού θα ανακαλύψει αυτό το ρηξικέλευθο το οποίο θα ανατρέψει τα όσα γνωρίζουμε για τον κόσμο όπως υπάρχει σήμερα. Ξέρω ότι οι μελέτες για τον εγκέφαλο είναι πολύ δημοφιλείς και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πολύ δαπανηρή, πολύ περίπλοκη, αλλά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να βρούμε τι είναι μέσα στο κεφάλι μας. Πάρα πολύ ωραία αυτά και βλέπω μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Και επίσης να συμφωνήσω και με τους συναδέλφους που μίλησαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μικρές μεν αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά μπορούν να είναι ιδιαίτερα καινοτόμε. Εγώ συμμετείχα σε κάποια καλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέδειξαν ότι πολλές καινοτομίες μπορούν να προέρθουν από αυτές τις μικρές μονάδες. Να τους ε, βοηθήσουμε λοιπόν, διότι πέραν από την έρευνα και την καινοτομία μπορούν να εργαστούν, οι άνθρωποι είναι πιο ικανοποιημένοι, είναι αυτόνομοι, μπορούν να προσφέρουν και να οικοδομήσουμε μια νέα Ευρώπη. Κάτι ακόμα. Να σας πω ότι επειδή εγώ εκπροσωπώ τις κοινωνικές επιστήμες, ε, θεωρώ ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε άλλες επιστήμες. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ο συνάδελφος ο καθηγητής Πρόντι, παρά το γεγονός ότι αυτός είναι εκπρόσωπος της ε, αμυγούς επιστήμης. Ε, μας επέστησε την προσοχή και στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές πτυχές και τον ευχαριστώ πολύ, περιμένω περισσότερα. Να συνοψίσω τώρα. Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι ένας χώρος ευτυχισμένων ανθρώπων, η κοινωνική και ψυχολογική έρευνα δεν θα πρέπει να παραγωνιστεί. Παραδείγματος χάρη, το άγχος. Δύο λόγια επιτρέψτε μου να πω ακόμα. Υπάρχει μια μελέτη για το άγχος στη Γερμανία. Γιατί ασχολούνται αυτοί και όχι εμεί. Και τέλος, μια τελευταία ερώτηση είναι δική σα αρμοδιότητα. Ίσως Πώς ε, χαρτογραφείται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ε, με ανθρώπους οι οποίοι θα αξιολογήσουν τα διάφορα προγράμματα. Σας παρακαλώ να τηρείτε λίγο περισσότερο το χρονοδιάγραμμα και για τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί τελείως δεν θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Γέρικ. Kiedy mowa o procedurach i o poszanowaniu uczciwych zasad gry, to uważam, że podstawą byłaby anonimowość προέκτου. A dlaczego? Bo wielkie znane firmy... ευχαριστώ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι για την ανωνυμία κάποιων τέτοιων έργων, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες τεράστιες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως ε, χωρίς την ανωνυμία τους χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλα πιο μικρά έργα. Για παράδειγμα, στην Πολωνία. Ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει να μπλοκάρονται κάποια έργα τα οποία θεωρούνται από κάποιου ω επικίνδυνα. Γιατί λοιπόν δεν αποφασίζουμε να ε, ανωνυμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα έργα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή και επιτρέψτε μου ε, ε, κάποιες παρατηρήσεις καταρχάς για τις πιστώσεις πληρωμών. Εμένα με εκπλήσει, διότι όταν δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου είπε ότι δεν θα υπογράψω ποτέ εάν δεν είναι καλυμμένες και πιστώσεις υποχρεώσεων. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε λίγο αυτή την πληροφορία. Ευχαριστούμε για όσα έχετε κάνει για την απλοποίηση. Η ερώτησή μου είναι πώς βλέπετε το μέλλον σε σχέση με την κατάσταση που μας παρουσιάσατε. Στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχει και μια ρήτρα πολιτικής αναθεώρησης το 2016, διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά νέα πολιτικά στοιχεία, τα κράτη-μέλη θα ισορροπήσουν ίσως τα δημόσια οικονομικά τους, ε, ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο να μην ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Κοινοβούλιο, ένα νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μήπως θεωρείτε ότι λόγω της συζήτησης που θα γίνει για τις ευρωεκλογές του 2014 θα μπορούσαμε ίσως να δοκιμάσουμε και αυτή την ιδέα η πολιτική έρευνας να είναι μια νέα κοινοτική πολιτική όπως κάναμε και με τη Γεωργία. Οι ε, εθνικές ε, ε, πιστώσεις πέρασαν σε κοινοτικό προπολογισμό και υπάρχει ένα κοινό όραμα. Και τέλος, πώς βλέπετε το συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Εγώ είχα ζητήσει να γίνει έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο αλλά και από τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε έλεγχο σε τρία επίπεδα, περιφέρειες, έθνη, Ευρώπη, για παράδειγμα, σε θέματα άμυνας έχουμε 27-28 στρατούς, ε, υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν έχουμε τίποτα κοινό και δεν έχουμε ούτε καν ένα κοινό φωτοτυπικό και υπάρχει και το θέμα της έρευνας. Γιατί λοιπόν να μην ε, τεθεί το θέμα της έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Φαν Ρόμπαϊ θα μπορούσε ίσως να ε, ρωτήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για θέματα όπως η άμυνα και ε, πραγματικά εμένα με εκπλήσει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2014 όταν ε, συζητούσαμε το θέμα του ορίζοντα 2020 το 2011-2012 και συμφωνήθηκε να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα της διαδρομής, θα τα συζητήσει. Δύο λόγια κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, εξετάσει την ανταγωνιστικότητα, το κόστος της ενέργειας, ε, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τις υποδομές, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αναφερόμαστε και στην ευηή ανάπτυξη και στις γενικές τεχνολογίες. Δεν υπάρχει συνολικό όραμα για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως ήγηκε η ώρα να εισαγάγουμε και αυτή την έννοια και να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική της επιστήμης και της έρευνας. Ευχαριστώ. Κορέρα Ντεκάμπο. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσά, κύριε Γενική Διευθυντά που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Στις δηλώσεις σας για τις συμφωνίες ε, ε, που μας απασχολούν σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ισότητα των φύλων, κοινωνικές επιστήμες ε, και το καθεξής περιορισμός της γραφειοκρατίας και το Ευρωπαϊκό ξέρετε, Συμβουλίο Έρευνα. Όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερως. Έχω και κάποιες ερωτήσεις όμως να σας κάνω. Είναι σαφές και η εισαγωγή σας ήταν ιδιαίτερως ευρεία. Οι απαντήσεις σας είναι πιο ενδιαφέρουσες γιατί είναι πιο συγκεκριμένες. Αυτό είναι λογικό. Δύο ερωτήσεις λοιπόν έχω να σας κάνω. προς το τέλος του τελευταίου προγράμματος έγινε λόγος για την εθνική χρηματοδότηση και τα εθνικά μέσα. Μας φαίνεται ότι λοιπόν αυτά πλέον τερματίζονται με το 7 πρόγραμμα πλαίσιο θα είναι δυνατόν να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση από πλευράς της Ένωσης ε, για τα περιφερειακά θέματα, περιφερειακά κονδύλια. Ο κ. Γιώχανσον το ανέφερε το θέμα αυτό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Γενικής Διεύθυνσης σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Ένα άλλο θέμα. Ε, γίνεται μια επένδυση σε αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο. Μήπως όμως έτσι περιορίζουμε κάπως τις ερευνές μας υπάρχουν και γίνονται τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες. Χθες ε, έγινε ένα εργαστήριο για τις χημικές διεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποθήκευση της ενέργειας. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο φοβάμαι ότι είμαστε κάπως ξεκαπερασμένοι. Δεν ξέρω αν τα αυτοκίνητα υδρογόνου είναι πιο καλά, πιο κακά από τα ηλεκτροκίνητα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να υποστηρίξουμε ή το ένα ή το άλλο σε ό,τι αφορά τώρα τις ασθένειες αυτές. Ίσως εδώ θα ήταν χρήσιμο και ενδιαφέρον να καταστρωθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα φάρμακα αυτά, τα οποία διερευνώνται περιορισμένα Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια χρηματοδότηση από πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά κάποιου συγκεκριμένου ασθενεί και υπάρχουν τέτοια ζητήματα για τι ασθένειε αυτέ. Και όντω θα μπορούσαμε να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ. Είπαμε πολλές φορές ότι τα αποτελέσματα από αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο είναι δυνατόν ε, να αποτελέσουν ένα ορόσημο για ε, την προϊστορία και την ιστορία των πραγμάτων Το πιο σημαντικό είναι πώς θα γίνει η απλούστευση, πώς θα γίνει η απλούστευση όσον αφορά τη συμμετοχή. Παραδοσιακά έχουμε εκεί πέρα ε, παράπονα, καταγγελίες από τους ερευνητές, από τις ΜΜΕ, από τα πανεπιστήμια. Είναι, είναι, είναι πάγιο το πρόβλημα εκεί πέρα. Έχω και εγώ προσωπική εμπειρία. Επομένω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια που έχει τα μέσα προ τούτο, να δει πώ θα μπορέσει να εποπτεύσει, πώ θα μπορέσει να υπάρχει μια εποπτεία, να ξεπεράσουμε τους φραγμούς και κατά τον τρόπο να μπορέσει να οριοθετήσει το πριν από το μετά. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις. Να φτάσουμε στο ποιοτικό άλμα αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με τα προγράμματα πλαίσιο. Πιλάρ, σε ευχαριστούμε. Ο Χόκμαρκ, έχω δύο σύντομε ερωτήσει να κάνω. Καταρχά, είναι στόχος εδώ και καιρό του Κοινοβουλίου, αλλά και όλων μας, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα προγράμματα πλαισίου. Και επίσης ε, υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί το πώς θα δαπανούνται οι πόροι. Ελπίζω η απόφαση που πήραμε να συνάδει με την ε, μείωση της γραφειοκρατίας. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, αλλά και το τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι οι ερευνητέ σε όλη την Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν λιγότερη γραφειοκρατία όταν ε, χρησιμοποιούν τα προγράμματα αυτά. Δεύτερη ερώτηση, η οποία ήδη έχει τεθεί για τις ευκαιρίες που συνδέονται. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σχέδιο ε, πλαίσιο για τα διαφορετικά ταμεία. Πώς ε, λοιπόν θέλετε να διευκολύνετε την πρόσβαση σε αυτά. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Πρόεδρο ότι ήμουν πάρα πολύ σύντομο στι ερωτήσει που έθεσα. Συνάδελφο Ήμπνερ, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πάρα πολύ θετικό το ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 πρόκειται να έχει επιπτώσεις πολύ θετικές. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενικέ για την ενημέρωση. Πρόκειται να ανοίξετε νέους δρόμους για τις ΜΜΕ. Γιατί οι ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την καινοτομία και για την απασχόληση. Αφού λοιπόν θα καλύψετε με της ΜΜΕ από αυτήν την ειδική υπηρεσία θα πετύχουμε κάτι σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό να απλουστεύσουμε τις σχετικές διαδικασίες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και έτσι οι ΜΜΕ να μπορέσουν να προστατολιστούν προς την καινοτομία χωρίς πρόβλημα. Επίσης είναι σημαντικό να δώσουν προτεραιότητα στον ενεργειακό τομέα και να έχουμε 15% αύξηση για την ενέργεια σα ερωτώ όμως, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δεν θα ήταν σωστό να καλύψουμε διάφορα κέντρα αριστείας στην Ευρώπη, να προσφέρουμε εκεί υποτροφίες και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε απαντήσεις για τις νέες τεχνολογίες και την αποθήκευση ε, των νέων μορφών ενεργείας. Γιατί υπάρχουν νέες μορφές ενεργείας, αλλά δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε ε, όταν χρειάζεται. Άρα, να έχουμε πετύχει κάτι μέχρι το 2030, να κάνουμε επομένω νέες προσπάθειες, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις νέες μορφές ενέργειας. Και έτσι τελικά να βρεθούμε ε, στην ευχαριστήση να έχουμε αξιοποιήσει τα χρήματα που υπάρχουν. Ευχαριστούμε την κυρία Χίπνερ. Τελείωσαν οι ομιλητέ. Ο κύριο ε, Σμιτ έχει το λόγο. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε Σαρτόρη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα διάφορα σχόλια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη να συζητήσετε. Αναφέρθηκε με σαφήνεια από την ε, πρώτη παρέμβαση του Πολωνού Ευρωβουλευτέ ότι θα πρέπει να προβλήψουμε ε, στον ορίζοντα 2020 ε, διαφορετική βασική έρευνα και ασφαλώς αυτός είναι ο στόχος του ERC. Δεν έχουμε στον ορίζοντα 2020 μόνο εφαρμοσμένες ε, έρευνες. Υπάρχει ένα, μια μεγάλη πρόβλεψη για διερευνητική έρευνα τέτοια και μελέτη. Αναφέρεται τη χαρτογράφηση του κεφάλου. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα προγράμματα δισεκατομμύριων ευρώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο το διαχειρίζονται οι συνάδελφοι από το DigiConnect. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, γιατί ο Γέφαλος ασφαλώς είναι μια ε, απροσπέλαστη περιοχή, στην οποία πολλά πρέπει ακόμα να ανακαλύψουμε, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή με τις νέες ασθένειες που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο τα τεχνικά ζητήματα, οι φυσικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες, αλλά και κοινωνικά, οικονομικα θέματα έρευνας. Στην προσέγγιση μας θα θέλαμε οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, είτε σε ό,τι αφορά θέματα ε, ασθενειών, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, οι συμπεριφορικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να συμπεριληφθούν, γιατί μιλώντας για ένα φαινόμενο όπως το διαβήτης για παράδειγμα, το θέμα δεν είναι μόνο να αναπτυχθούν νέα φάρμακα, είναι και θέματα συμπεριφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να ενταχθούν και αυτές οι διαστάσεις, ε, οι κοινωνικές, οι ανθρωπολογικές, στην στο πρόγραμμα αυτά, στα αυτά. Ένα ενδιαφέρον σχόλιο έγινε για την ανωνυμία των έργων. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό, είναι η ανωνυμία της διαδικασίας αξιολόγησης και των υπευθύνων αξιολόγησης, γιατί φαντάζεστε αν είναι κανείς ε, υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενός έργου 50 δισεκατομμυρίων και το απορρίψει, δεν έχει πολύ μεγάλο μέλλον πλέον το συγκεκριμένο άτομο αν αποκαλυφθεί ότι αυτός το απέρριψε το πρόγραμμα. Να μην δημοσιεύονται λοιπόν τα ονόματα τα μεμονωμένα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος του αξιολογητή σε αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, κύριε Οντή, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και θα σας δώσω και γραπτά αν θέλετε κάποια στατιστικά στοιχεία. Στην παρούσα φάση έχουμε έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις πληρωμές αυτές και χρησιμοποιούμε αυτή την προχρηματοδότηση. Περιορίζουμε τις ενδιάμεσες πληρωμές, αλλά δημιουργούμε και ένα σύνδεσμο με τις πιστώσεις πληρωμών που θα χρειαστούμε κάποια στιγμή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ε, μία παράδοση έλλειψης ε, πιστώσεων πληρωμών και παράλληλα χρειάζονται και πληρωμές για προχρηματοδότηση για τον ορίζοντα 2020 και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν τελικά σε αδιέξοδο σε ένα-δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν την βοήθειά σας να αναζητήσουμε σχετικές λύσεις. Μας παρουσιάσετε μια ενδιαφέρουσα ιδέα σε ό,τι αφορά την επιστήμη και την κοινοτομία και την τοποθέτησή του στο κέντρο της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και το θέτει πάντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς από πλευρά μας ασφαλώς και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι. Αναφέρθηκα και στην πρωτοβουλία αυτή με τον Αντιπρόεδρο Ρεν. Και σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση τη επιστήμη και τη ε, καινοτομία στην κορυφή των προτεραιότητων μα, των πολιτικών προτεραιότητων μα. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό ακόμα. Πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα προτού ε, η έρευνα και η καινοτομία τεθούν ω συγκεκριμένε συστάσει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα εργαστούμε λοιπόν και άλλο προ την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε βαθμία να το προσεγγίσουμε το στόχο αυτό. Αρκετοί εξημών αναφερθήκατε στο σύνδεσμο με τα διευθυντικά ταμεία. Με την συνεργασία με τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο διασφαλίζουμε ότι οι εταιρικέ σχέσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα των κριτών μελών λαμβάνουν υπόψη την επιστήμη και την καινοτομία. Με ευφύ τρόπο, όχι μόνο επειδή δηλαδή είναι στη μόδα να υπάρχει ένα κέντρο νανοτεχνολογίας να χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο τα κονδύλια αυτά. Όχι, θα πρέπει να δαπανώνται σκόπιμα. Αναφέρθηκε από διάφορους βουλευτές το θέμα του ηλεκτρισμού, της ενέργειας, της αποθήκευσης που αποτελεί θέμα κλειδί, πρόβλημα. Εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Ελπίζουμε και αυτή η ιατρική σχέση για τις ε, κυψέλες αποθήκευσης υδρογόνου να αποτελέσει μια λύση, γιατί το θέμα αυτό μας εμποδίζει πολύ. Αναφέρθηκαν και αυτές οι ασθένειες, σπάνιες ασθένειες, οι πολύ σπάνιες ασθένειες. Δημιουργήθηκε πρόσφατα ένα σχετικό δίκτυο για αυτές τις πολύ σπάνιες ασθένειες με το Εθνικό Ινστιτούτο, τι τον είπα, του Καναδά της Ιαπωνίας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό το θέμα των πολύ σπάνιων ασθενειών και της σχετικής και απαραίτητης ε, ε, των σχετικών φαρμάκων. Μιλήσατε κυρία Πιλαρδικαστήγιο για τα θέματα πρόσβασης, ότι ο κόσμος θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στα προγράμματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες για τα προγράμματα διατίθενται online στο διαδικτύο με τρόπο φιλικό προς το χρήστη. Τι είναι όμω σημαντικό σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν καλά σημεία επαφή. Και αυτό το τονίζουμε διαρκώ. Γιατί η Γενική Διεύθυνση Έρευνα δεν είναι δυνατόν να πάει σε όλε τι περιφέρειε, σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Αυτό θα πρέπει να γίνει από καλά σημεία επαφή, τα οποία ορίζονται από τι εθνικέ αρχέ, τα οποία εμεί εκπαιδεύουμε και τα οποία εμεί πιστοποιούμε προκειμένου να είναι υψηλή ποιότητα. Αλλά αυτό το θέμα τη προσβασιμότητα, ιδιαίτερα για του καινούριου φορεί, είναι πολύ σημαντική. Να μην περιοριζόμαστε δηλαδή στους ίδιους φορείς. Εθνικά σημεία επαφή λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά. Άρκετοι συνάδελφοι έθεσαν ερωτήματα για την ε, γραφειοκρατία και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό με τη μέτρα. Πολύ απλό, κυρία Καρβάλιο. Ε, έχετε καταρτήσει μια έκθεση με 52-54 δράσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. μπορώ να σας αναφέρω ένα προς ένα τα στοιχεία αυτά. Το έγγραφο αυτό λοιπόν εγκρίθηκε από την Επιτροπή αυτή και αυτό αποτελεί το leitmotiv μας, αν θέλετε, τον απότερο στόχο μας για την ε, ατζέντα της απλοποίησης. Και νομίζω ότι πολλά από τα συγκεκριμένα μέτρα καταφέραμε να τα εντάξουμε στους ε, κανόνες για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς Νομίζω λοιπόν ότι από αυτήν την άποψη πετύχαμε πολλά. Και τα τελευταία σχόλια είχαν να κάνουν για, με τον προπολογισμό και την αύξηση του προπολογισμού για την ενέργεια. Και αυτό λοιπόν είναι στόχος μας σε ό,τι αφορά τα θέματα αποθήκευσης. Ελπίζουμε σύντομα να δούμε στην πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο θέμα αυτό. Ζητούμε την υποστήριξή σας για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά το πακέτο για τις συμπράξεις αυτές. Νομίζω στις 19 Φεβρουαρίου έγινε, θα προβλέπετε μάλλον ο τελευταίος τριμερής διάλογος. Θα είναι σημαντικό όμως να πετύχουμε συμφωνία τότε. Ελπίζω λοιπόν αυτό να εγκριθεί σύντομα. Και τέλος θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες όχι μόνο προς εσάς, αλλά και από τους συναδέλφους μας που είναι εδώ στην αίθουσα, οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ είναι εξαιρετικοί και η δουλειά του ήταν εξαιρετική σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Horizon 2020. Ευχαριστούμε εξ ονόματο της Επιτροπής μας τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σμιτ. Να σα ευχηθούμε καλή δουλειά και στο επανειδήν. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Γι' αυτό λοιπόν όσοι θέλουν να αποχωρήσουν παρακαλώ ησύχως. Και να περάσουμε στην δημόσια κρόαση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. που σχετίζεται και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το ορίζοντα 2020.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 seconda parte della mattinata. Siamo un Ξεκινούμε το δεύτερο τμήμα της ημέρας. Ε, έχουμε καθυστερήσει λίγο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας ε, για ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας και σχετίζεται με τον ορίζοντα 2020 τους στόχους ε, οι οποίοι αναφέρθηκαν ε, ιδιαίτερα σήμερα το πρωί στη συζήτηση, το πώς ε, δηλαδή θα υλοποιήσουμε αυτές τις δύσκολες και περίπλοκες προπτικές, να θέσουμε εντός του 2014 τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Για το θέμα αυτό, για το οποίο υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες τους τελευταίους μήνες ε, και κατά την άποψή μας υπάρχει αφενός η ανάγκη αλλά και η πολιτική ανάγκη να καταλήξουμε σύντομα σε αυτούς τους στόχους. Να δώσω λοιπόν καταρχώς το λόγο στον ε, Jean-Pierre Bourguignon, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας. Παρακαλώ κύριε Bourguignon. Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, euh, je suis euh, très... Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, με μεγάλη μου τιμή που εμφανίζομαι εδώ να σα μιλήσω μετά την έλευση των καθηκόντων μου, να θίξω κάποια θέματα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα ή ERC. Αποτελεί την υλοποίηση των δυνατοτήτων της Ένωσης χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους ε, θεσμικά ιδρύματα και θεσμούς. Ε, αυτό έγινε ε, επί τη βάση μιας πρωτοβουλίας για την επιστήμη, διάφορα υπουργεία, κρατών μελών και ο Επίτροπος Μπισκέ, ο οποίος μετέπειτα έγινε συνάδελφός σας, βοήθησαν στη δημιουργία της υπηρεσίας μας και και ο Ποτότσινο και επίσης ως Επίτροπος βοήθησε και επίσης εντάχθηκε και στην πρωτοβουλία ιδείας ε, του 7ου προγράμματος πλαισίου. Φυσικό ήταν να ασχοληθεί ο Γενικός Διευθυντής Σμίτσα και η Επιτροπός ε, Κουίν ε, να αποτελέσουν ένα από τα θέματα αναφοράς του προγράμματος Horizon 2020 και εσείς ασχολείστε, έχετε φροντίσει για την πρικοδότησή μας. Όπως γνωρίζετε βάσει του Horizon 2020, το ERC σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο έχει διπλασιάσει την πρικοδότησή του. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εξέλιξη του Ιδρύματος. Οπότε αυτό δεν αποτέλεσε φυσικά παρά μια ενθάρρυνση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και ίσως ε, θα έχουμε επέκταση αρμοδιοτήτων μας περί τα τέλη του προγράμματος ορίζων. Ήταν η υποδοχή ενθουσιώδης από την επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Τα δευραβεία που έχουμε απονείμει χαιρετίστηκαν από όλες τις χώρες. Τώρα, όσον αφορά το βασικό ερώτημα. Εάν καλύπτουμε κάποια βασικά προγράμματα, οπότε βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα σημαντικό μείγμα καινοτομία και έρευνα στο έργο μας. Βλέπουμε ότι οι χώρες και οι περιφέρειες που τα πάνε καλύτερα Έχω στο πάνε καλύτερα και στην έρευνα. Η βασική έρευνα επομένως βοηθάει πολύ, οδηγεί σε διπλωματούχους και ερευνητές υψηλού επίπεδου, οι οποίοι εμπλέκονται σε κάποια προγράμματα τελείως ανοιχτά. Οπότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προσδόκητα σε διαφορετικούς τομείς, σε κάποιες εκπλήξεις, γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ καλή προετοιμασία για να αποφύγουμε κάποιο είδου προβλήματα και βραχικυκλώματα. Οπότε βλέπουμε τι έγινε με την εταιρεία Google. Δύο μαθηματικοί βρήκαν έναν αλγόριθμο, τελείως νέο. Τώρα το χρησιμοποιούν μαθηματικοί για διάφορες αποδείξεις και ήταν πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίε για ένα οικονομικό μοντέλο και δημιούργησαν αυτή την εταιρεία. Την εταιρεία που την ξέρουμε σήμερα ως Google ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλοι συνέχεια χρησιμοποιούν το Google. Δεν πληρώνουμε. Κάποιοι βέβαια πληρώνουν. Έτσι υπάρχει και είναι τόσο ε, ακμάζουσα αυτή η εταιρεία. Ήταν καταρχήν απλό, αλλά αξίζει να το αναλύσει κανείς το φαινόμενο. Πώς λοιπόν έχουμε μια σύγχρονη επιστημονική προσπάθεια που κατόπιν μεταφράστηκε σε τόσο σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Άλλο παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι μια βιομηχανική πρωτοβουλία στην ΕΛΒ ένας μηχανικός βρήκε ένα πάρα πολύ εξύπνο τρόπο να κωδικοποιήσει το σήμα όσον αφορά το, το, το, το πετρέλαιο και την έρευνα και τελικά βρήκε ένα καινούριο τρόπο να επεξεργάζεται το σήμα. Και η εφαρμογή τελικά δεν ήταν η έρευνα σχέση με το πετρέλαιο, αλλά αυτό χρησιμεύσε και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς σαν ανάλυση σήματος, εικόνας, ήχου. Έγινε επομένως ένα μέσο πάρα πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση της ε, εικόνας και είχε να κάνει επίσης και με την ανάπτυξη του πρότυπου ή του πρωτοκόλου JPEG 2000. Να, ένα απλό παράδειγμα. Όπου είχαμε μια ανακάλυψη από μηχανικό, είχαμε εμβάθυνση από θεωρητικούς, μαθηματικούς, ε, κομπιουτεράδες, τέλος πάντων είδαμε πώς διευρύνθηκε μία ανακάλυψη για να γίνει ένα εργαλείο γενικευμένης χρησιμότητας. Έτσι λοιπόν είδαμε πώς συνδυάζεται ο ένας κλάδος με τον άλλο. Κάτι άλλο τώρα. Να σας πω ότι το Συμβούλιο Έρευνας έκανε την επιλογή να αφιερώσει τα δύο τρίτα της προκοδοτησής του στους νέους ερευνητές. Έχουμε τρία προγράμματα σήμερα. Starters, το πρώτο. Ένα άλλο Consolidators, δηλαδή ε, πρόκειται για κάποιους μεταξύ 7 και 12 ετών, καλύπτονται. Mm -hmm. Και επίσης, το τρίτο είναι για τους μεγαλύτερους. Κάναμε αυτή την επιλογή από το Συμβούλιο και κατανείμαμε τα δύο τρίτα των πιστωσιών μας. 1,7 δις ετησίως έχουμε. Και αυτά τα αφήνουμε επομένω στους νέους ερευνητέ για να του δώσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ομάδες τους. Να, ένα μήνυμα εμπιστοσύνη το οποίο στείλαμε. Σε σχέση με το ότι είμαστε αποφασισμένοι να πείσουμε ότι στην Ευρώπη μπορούμε να έχουμε ερευνητικές ομάδες. Και αυτό να διαρκέσει, να είναι βιώσιμο. Βέβαια, ε, πάρα πολλές χώρες διεκδικούν το, να κρατήσουν τους, ε, τους πιο λαμπρούς από αυτούς τους ερευνητές. Δεν κατακλείω τώρα να σταθώ σε δύο θέματα τα οποία έχουν ε, θυγεί από τους προλαλήσαντες σε σχέση με την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντού. Αλλά και εσείς τα θίξατε στις παρεμβάσεις σας. Πρόκειται για δύο ανισορροπίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Έρευνα, κάτι το οποίο αφορά την γεωγραφική κατανομή και κάτι που αφορά το, το πώς ελκύουμε τους ερευνητές. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε πώς θα έχουμε περισσότερο προσωπικό, περισσότερους ερευνητές, αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Η διαχείριση αυτού του προβλήματος δεν είναι τόσο εύκολη, θα πρέπει να τεθούν κάποιοι στόχοι, ήταν σαφής πάνω στους στόχους της Επιτροπής, ο κύριος Γενικός, και επομένως ε, τη κάθε επιστήμης είναι διαφορετική. Ε, εγώ είμαι μαθηματικός και εκεί δεν εκπροσωπείται πάρα πολύ καλά το αδύνατο φύλλο επειδή σε ορισμένε χώρες υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή, ε, αλλού είμαστε κοντά στην ισομερή συμμετοχή και οπότε έχουμε κάποιες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί που δεν είναι ομοιόμορφες αλλά είναι καλά στοχευμένες και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά κάποιου φραγμού ε, οι οποίοι δεν είναι τόσο χειροπιαστοί και αποθαρρύνουν τι γυναίκε. Κάτι άλλο που αφορά την γεωγραφική κατανομική ανισορροπία. Πρόκειται κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την αρμονική ανάπτυξη τη Ευρώπη. Γιατί πάρα πολύ συχνά σε χώρε που δεν έχουν ε, υποδομέ ε, εκεί υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης οπότε ε, υπάρχουν κάποιοι εξαίοντες ερευνητές οι οποίοι ε, δεν, προέρχονται από, από διαφορετικές χώρες από αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και είχαμε τη συνεδρία τη περασμένη εβδομάδα και αποφασίσαμε να είμαστε πιο δυναμικοί, ενεργητικοί σε αυτό και να προσπαθήσουμε να πλαισιώσουμε τέτοιε προσπάθειε για να αξιοποιήσουμε του πόρου των ε, διαρκτικών ταμείων, τόσο ώστε οι ερευνητέ από κάποιε χώρε όπου είναι λιγότερο αναπτυγμένες υποδομέ να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής ε, Διεύθυνσης, Περιφερειακής Πολιτικής μάλλον. Οπότε και το Συμβουλίο μας θεωρεί ότι μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαμόρφωση νέων εργαλείων που μπορούν να λειτουργήσουν. Θέλουμε οπότε έτσι να πλαισιώσουμε κάποιους νέους ερευνητές οι οποίοι παρά το δεν έχουν πάρει υποτροφία από μας έχουν ήδη επιλογή σε, σε, πρώτη φάση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον των χωρών τους. Ε, Ευχαριστούμε τον Ζαμπιαμπουργινιό. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, Ντέτλερ Μίλλερ Βίσνερ από την ομάδα της Airbus, ε, πρώην πρόεδρο του Διεθνές Συμβουλίου Αεροναυτικών Επιστημών. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Okay. Uh, could you make this operate Σα uh, uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Βιομηχανίας, αγαπητά μέχρι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω την ευκαιρία ως μόνος εκπρόσωπος της βιομηχανίας σήμερα να σας ε, παρουσιάσω τη δική μου μαρτυρία. Έχω κάποιες ερωτήσεις τις οποίες ε, θα σας ενδιαφέρουν ενδεχομένως γιατί έχουμε εκπροσώπους από τον επιστημονικό κλάδο και ίσως θα σας ενδιαφέρει να μάθετε που έχουμε έρευνα εκτός επιστημονικών ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τον όμιλο Airbus για τον οποίο εργάζομαι, θα βλέπετε στη διαφάνεια ότι εμείς από μόνο μας ε, δραστηριοποιούμεθα με 5.000 άτομα στην έρευνα. Μιλώντας λοιπόν για επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας, η έρευνα έχουμε 5.000 ε, άτομα σε τέτοια θέματα, σε τέτοιου τομεί τεχνολογίας που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την έρευνα. 3% του εργατικού μας δυναμικού περίπου. Σε σύγκριση λοιπόν αυτό με μια χώρα σε ό,τι αφορά και τον κύκλο εργασιών μας, ε, θεωρώ ότι, έχουμε, ότι πληρούμε του όρους της Ευρώπης. 3% το αξιοποιούμε στην ερεύνα και η υποστήριξη από πλευράς ε, τέτοιων ε, μάλλον είναι το 1 τρίτο του ερευνητικού μας ε, προπολογισμού σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, σε άλλες βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία, Είμαστε λοιπόν πιο εντατικοί. Και μιλάμε λοιπόν για τη δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να σας πω ότι έχουμε ένα ε, ιδιαίτερο ταμείο, ένα ταμείο καινοτομίας, όπου χρηματοδοτούμε οι ιδέες που έχουν να κάνουν με τέτοια θέματα αεροναυτικής για νέες επιχειρήσεις. Πέρσι λοιπόν είδα και βρήκα δύο επιχειρήσεις με επιχειρήσεις για έναν ανείχνευτη νερού, όπου γίνεται ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων του πόσιμου νερού μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και η άλλη εταιρεία από πλευρά ε, βιομηχανίας ε, και εταιρεία ε, κατασκευαστικής για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους παρόχους μας. Και θα επανέλθω λοιπόν σε τέτοια θέματα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα από τους μεγαλύτερους φακέλους IP στον κόσμο. και κοιτώντα και τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε ε, στο scoreboard στις κορυφαίες 50 εταιρείε του κόσμου, ίσως και στις κορυφαίες 30. Με τα μέτρα λοιπόν αυτά για τη μεταφορά IP για τους ε, ε, παρόχους και στις επιχειρήσεις μας, ουσιαστικά διαδίδουμε τα αποτελέσματα της έρευνας από το δικό μας τομέα τον οικονομικό κλάδο και συνδράμουμε και εμείς την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων ε, βιομηχανικών κλάδων και κυρίως τον κατασκευαστικό κλάδο. Να κοιτάξω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα ποια είναι η σχέση μας με τις μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η έρευνα στο ιστορικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, και εγώ να σας πω για το δικό μας το κλάδο, η καλύτερη συμβολή για την επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η συνεργασία τους με την ΕΑΜΣ. Γιατί η στρατηγική ανάπτυξη ενός αεροσκάφους δεν αναπτύσσεται από τους μεμονωμένους παρόχους. Πρόκειται για πολύ συγκεκριμένες αγορές. Εμείς λοιπόν οι e χρειαζόμαστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας χρειάζονται. Γιατί τις χρειαζόμαστε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της ε, υψηλής δραστηριότητάς της. Ε, είμαστε λοιπόν μια, ε, ένας κλάδος με 5.000 ερευνητές και είμαστε λοιπόν σαν την ε, Ευρώπη σε ό,τι αφορά την παροχή τέτοιων κονδυλίων. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, είναι δύσκολη η λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μας είναι ένας τρόπος να λαμβάνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις. Ο διευθυντής για παράδειγμα μπορεί να αποφασίσει πολύ πιο γρήγορα κάτι σε σχέση με, μια μεγάλη, με ένα μεγάλο όμιλο. Από την άλλη το πλανέκτημά μας είναι ότι λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο λήψη αποφάσεων στο παγκόσμιο, στο παγκόσμιο προσκήνιο, στην παγκόσμια αγορά. Και πάλι να επανέλθω στο θέμα του IP, γιατί συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν τα απαραίτητα για τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησίας IP αν συνεργαστούν με μεγάλους ομίλους, είναι συνειδιοκτήτες των διανετικών δικαιωμάτων αυτών και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε έτσι να προωθούμε τη γνώση στο εσωτερικό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε όμως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να υποστηρίξουμε γιατί οι ε, γενικές γραμμές δεν δέπανουν πολλά στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τις μπλέκουμε με έναν έξυπνο τρόπο στην ε, έρευνα για την ανάπτυξη. Τώρα, τι περιμένουμε από την πολιτική για την έρευνα στην οριστό 2020. Στο Clean Sky 2, στο Caesar, στο ηλεκτρονικό GTI XL και σε άλλα προγράμματα, ακόμα και σε θέματα ασφάλειας, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός για να ε, συνάδουμε στην αγορά με τις προδιαγραφές του ΠΟΕ και έτσι με τον τρόπο αυτό να φέρουμε χρήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, λανσάρντας σε έγκυρο χρονικό σημείο προϊόντα τα οποία θα κάνουν την Ευρώπη ανταγωνιστική. Και έτσι λοιπόν έχουμε και θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προωθούν την κοινοτομία. Από την άλλη χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία έρευνας όπως αυτά. Δεν είμαστε πεπισμένοι όμως ότι η αύξηση των project ε, έρευνας επίπεδου 2 είναι απαραίτητα προς το όφελος της ε, ανάπτυξης αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοια στοιχεία, χρειαζόμαστε συνεργασία με τη Γερμανία, χρειαζόμαστε και ξέρουμε τι λαμβάνουμε από τα κέντρα έρευνας. Τελευταίο σημείο, τι περιμένουμε από τον ορίζοντα 2020 συγκεκριμένα. Κατά κάποιο τρόπο, σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι με τους ε, κανόνες για τη συμμετοχή και έχουν γίνει συζητήσεις με τα κρατημέλη, με την Επιτροπή για το άρθρο 46.3 σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τη συμμετοχή. Χαιρόμαστε που το άρθρο αυτό πλέον έχει διαγραφεί από τον κανονισμό αυτό, γιατί αναφέρει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να παρουσιάζει όλο το σύνολο των γνώσεων σε ό,τι αφορά τα διανετικά δικαιώματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για μελλοντικέ χρήσεις. Αυτό λοιπόν θα σκότωνε την βιομηχανία, αν δίναμε δηλαδή την ελεύθερη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει συμφωνία Grant σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ακούσαμε και θέματα ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αν θα πρέπει να δημοσιεύσω όλα μου τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην κυβερνοχώρο, τα δίνω κατευθείαν και στους hacker. Λυπάμαι. Λοιπόν, η διαγραφή του άρθρου 46 είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζουμε έτσι να παραμείνει. Και τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πάθος μου για τα αεροσκάφη. Σε ό,τι αφορά το Flight Path 2050 για την ε, βελτίωση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Αυτό είναι προσωπικός μου στόχος, γιατί από την αρχή του, του Φεβρουαρίου είμαι επικεφαλής ενός προγράμματος του ΙΦΑΝ για την χρήση σε 20 χρόνια ηλεκτρικών, ηλεκτροκίνητων ε, οχημάτων. Και θα δείτε λοιπόν τρία αεροσκάφη εδώ στην διαφάνεια, τα οποία λειτουργούν, πετάν με ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι λοιπόν το μέλλον. Ακούσαμε λοιπόν ότι γίνεται έρευνα για τις μπαταρίες κτλ. Εμείς είμαστε λοιπόν κατεξοχήν εταίρος για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά και τη σχέση με τις ηλεκτρικές μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα αυτοκίνητα. Είμαι πεπισμένος ότι εκεί είναι το μέλλον και για τα αεροσκάφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και φυσικά θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον καθηγητή εμέριτος Κάρλος Σαλέμα από το Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο της Πορτογαλίας. Παρακαλώ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Κύριε, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση πρόκειται να μιλήσω για τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά θα περιοριστώ στην ε, ε, πληροφορική και την επικοινωνία στο ICT που είναι ε, παρακλάδι του 7ου προγράμματος πλαίσιο και θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου ως εθνικός αντιπρόσωπος στα θέματα αυτά. Όλα τα συγκεκριμένα προγράμματα από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στις τηλεπικοινωνίες δηλαδή και στην τεχνολογία. Θα σταθώ σε έξι σημεία. Το πρώτο αφορά όπως και τα, ο δεύτερο και το τρίτο το τι και το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο το πώς. Πρέπει να πω ότι στις τηλεπικοινωνίες η Ευρώπη είχε ε, μια πάρα πολύ καλή έναρξη ε, διότι τα κινητά τηλέφωνα γεννήθηκαν στην Ευρώπη. Οι κινητές τεχνολογίες ε, ε, προέκυψαν από προηγούμενα ε, προγράμματα πλαίσιο, το τρίτο και το τέταρτο. Τώρα η Ευρώπη έχει χάσει τον ηγετικό της ρόλο στις κινητές, ε, στις τηλεπικοινωνίες, αλλά υπάρχει ελπίδα, υπάρχει το 5G το οποίο θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει τον διάδοχο του GSM και ε, τους χαμηλή χαμηλής ισχύω που πρέπει να υποστηριχθούν στο ονορίζοντα 2020 διότι είναι πολύ σημαντικό στις ε, προηγμένες τηλεπικοινωνίες και ίσως έτσι η Ευρώπη ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο. Αυτό πρώτο. Δεύτερον, τα πρότυπα για ε, οπτικοακουστικά, ε, για ηχητικά, για συμπίεση βίντεο, το MP3, το MPEG και την μετάδοση. Δυστυχώς και σε αυτά η Ευρώπη έχασε τον ηγετικό της ρόλο, παρά το γεγονός ότι υποστηρίχθηκαν από προηγούμενα προγράμματα. Το 7 πρόγραμμα πλαίσιο υποστήριξε προηγμένες τεχνολογίες ε, τρισδιάστατης τηλεόρασης που μπορεί να βοηθήσουν την Ευρώπη να ανακτήσει τον ηγετικό τους ρόλο, αλλά και γενικότερα να υπάρχουν περισσότερες συσκευέ στην αγορά. Χρειαζόμαστε όμως έγκριση κοινών προδιαγραμμών και νομικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Τώρα, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο. Οι οπτικές σύνε που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες προτάθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη και ο το πρώτο ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται ακόμα στην αιχμή των οπτικών ινών. Ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υποστήριξε καινοτόμε χρήσει των ε, επικοινωνιών μέσω οπτικών ινών, όπω για παράδειγμα το Radio Over Fiber και ε, θα πρέπει να συνεχίσει η υποστήριξη αυτών των επικοινωνιών μέσω φωτονίων και οπτικών ινών στον ορίζοντα 2020. Τώρα να περάσω σε ένα πιο ακαθόδε ζήτημα, το ποιος. Έχω βέβαια κάτι ακόμα να σας πω για το τι, το πώς θα διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο και να σας πω ότι το διαδίκτυο προκύψε από ε, ένα στρατιωτικό πρόγραμμα ε, και ε, οι επιστήμονες ε, μπόρεσαν να προχωρήσουν τις δραστηριότητες αυτές μέσω του προγράμματος πλαίσιο 6 και ίσως αυτό είναι το πιο μακρόπνο πρόγραμμα και θεωρώ ότι ορίζοντας 2020 θα πρέπει να υποστηρίξει προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου και σχετικές εφαρμογές. Και τώρα να περάσω στο πώς.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 Δυστυχώς τα προγράμματα του 7ου το προγράμματος πλαίσιο ε, θεωρούνται από τρίτους ως προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή ε, και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και το 2000, το, στον ορίζοντα 2020. Ε, μικρότεροι οργανισμοί, μικρότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να συμμετέχουν. Η συμμετοχή και ο συντονισμός σε μικρότερα προγράμματα είναι πολύ πιο εύκολη από μεγαλύτερα προγράμματα. Επομένως, τα μεγάλα προγράμματα δεν θα πρέπει να από τη μερίδα του λέοντος. Έχω δει επανειλημμένως ότι πολύ καλά μικρά προγράμματα δεν χρηματοδοτήθηκαν διότι ε, δόθηκε προτίμηση σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν τόσο καλό. Επομένως, η συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσιο είναι μια ε, δραστηριότητα η οποία προσφέρει και τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες. Όταν μειωθεί το κατώτατο όριο, τότε θα μπορέσει να υπάρχει και καλύτερη, μεγαλύτερη συμμετοχή και επομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους συμμετέχοντες να υποβάλουν υποψηφιότητες. Ε, πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με τους κανόνες απλοποίησης που εισήχθησαν στον ορίζοντα 2020. Όχι μόνο με τους κανόνες αλλά και τα κριτήρια επιλοξιμότητας ε, ε, που είναι ε, σημαντικά για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και ίσως το, όχι τόσο σημαντικό για επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το πρόγραμμα πλαίσιο εκφύσεως είναι περίπλοκο και υπάρχει και μεγάλη γραφειοκρατία, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα ε, με την απλοποίηση η οποία εισήχθη. Το μέσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι φαίνεται. Και έχω και τους ίδιους εφιάλτες που ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής ε, προηγουμένως, ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες. Είναι τόσο ελκυστικό αυτό το μέσο που ανησυχώ ότι μπορεί να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αποτελεσματικότητα. Means making Αποτελεσματικότητα μπορεί να σημαίνει περισσότερο ή και με, λιγότερα. Σημαίνει να έχουμε αποτελέσματα και όχι απλώς πολύ καλούς οικονομικούς ελέγχους. Η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν εντός του προπολογισμού μας ε, τα προγράμματα επιτυγχάνουν τους, ε, τις προδιαγραφές των στόχων. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνετε σε τεχνικούς ελέγχους και όχι σε οικονομικούς. Η οικονομική έλεγχη μπορεί να είναι ωραία και καλή, αλλά ε, μπορεί να μην είναι τίποτα ε, πίσω από όλα αυτά και πολλές φορές υπήρξαν απάτες στο παρελθόν που αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Τολμώ δεν να πω ότι παρά το γεγονό ότι είναι τολμηρή αυτή η δήλωση, οι οικονομικοί έλεγχοι θα πρέπει να πετούνται μόνο όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Μόνο τότε ε, θα πρέπει να ανησυχήσει κάποιο για τα παραδοτέα προϊόντα και να κάνει έναν οικονομικό έλεγχο για να διαπιστώσει τι συνέβη. Τέλος, η διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα κράτη-μέλη. Μέσω διαχειριστικών επιτροπών ε, του, δεν θα πρέπει να τους περιορίσουμε κι άλλο τις εξουσίες τους. Θα πρέπει να δίνονται έγκαιρες πληροφορίες στις ε, διαχειριστικές επιτροπές και πραγματικά αυτό δεν σας το λέω ελαφρά την καρδία. Θεωρώ ότι τα εθνικά σημεία επαφής ε, κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνίας στα οποία συμμετείχα ε, δεν έδινε πάντα έγινες πληροφορίες. Ε, πληροφορίες για τις ε, προτάσεις και τις υποβολές ε, στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς θα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει το κριτήριο με το οποίο αποφασίζουμε να είναι αριστεία και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, διότι οι δυνητικές συνέπειες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν και θα πρέπει... Ε, ότι ο Χέρτς που απέδειξε ότι ο Μάξουελ είχε δίκιο, όταν είπε ε, με τι κριτήρια το έκανε αυτό, είπε για κανένα λόγο, δε, με τίποτα. Μπορείτε να ζήσετε μόνο με κάτι το οποίο έχετε στη ε, στην τσέπη σας. Ε, τα κύματα λοιπόν που απέδειξε ο, Χέρτζ ότι ισχύουν βάσει του Μάξουελ δεν έχουν καμία αξία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ να προχωρήσουμε τώρα τις εργασίες μας. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σάσα Μπεζουχάνοβα, πρόεδρο της ομάδας υψηλού επίπεδου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία και πρόεδρο επίσης του Κέντρου Γυναικών στην Τεχνολογία στη Βουλγαρία. Παρακαλώ, η κυρία Σάσα Μπεζουχάνοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. όπως ανέφερε ο καθηγητής Bourguignon στην αρχή. Έχουμε δύο τομείς που θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουμε να είμαστε πρακτικοί για να εξελίξουμε και αναπτύξουμε την ερευνητική μας ε, επίδοση. Να έχουμε συνεργασία στους αντίστοιχους μηχανισμούς σε όλη την Ευρώπη για την έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερες γυναίκες. Θα πρέπει να τις ελκύσουμε στον ε, έρευνα. Θα προσπαθήσω αν όχι να δώσω λύση, τουλάχιστον να σας δώσω ευκαιρία προβληματισμού για το θέμα. αξιολογούμε το τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη για να είμαστε αποτελεσματικοί, για να είμαστε πρακτικοί. Για να μπορέσουμε να ελκύσουμε όχι μόνο αυτούς που ζουν στην Ευρώπη, αλλά κόσμο από όλο τον κόσμο. Και να δούμε επίσης την παγκόσμια συγκυρία. Τι γίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα καλύψουν όχι τις διοικητικές, αλλά όλες τις ανάγκες. Η κρίση άφησε πολύ κόσμο στην ανεργία. Έχουμε σήμερα περίπου 26.000 εκατομμύρια διορθώνει ομιλήτρια άνεργους στην Ευρώπη και το 60% αυτών είναι νέοι. Οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστούμε τον επιχειρηματικό κόσμο, πώς θα έχουμε και επιστατηγικές, τι ανάγκες έχουν οι επιχειρήσεις. Έχουμε κάποιες γιγαντιές εταιρείες που δεν είναι όμως τόσο αποτελεσματικές σήμερα. Άρα θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα βρούμε νέες ιδέες και νέους μηχανισμούς για την έρευνα. Και αυτά όλα να γίνουν γρήγορα. πώς στον επαγγελματικό χώρο θα υπάρχει αποτελεσματικότητα. Να δούμε τι γίνεται στην Ασία, στον Ελληνικό, στην Νότια Αμερική. Εκεί έχουμε νέους με δεξιότητες από την Ευρώπη, οι οποίοι εκεί βρίσκουν ευκαιρία για έρευνα, αλλά βρίσκουν και δουλειά σε αυτέ τι νέε αναδυόμενες περιοχές. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι αρκετά αποτελεσματική για να μπορέσει να τους προσφέρει μια σταδιοδρομία, μια δουλειά. Επίσης, αν αξιολογήσουμε την καινούργια, ε, το καινούργιο τοπίο, το γεωπολιτικό και οικονομικό, θα διαπιστώσουμε σαφώς ότι οι χώρες BRIC, η Κίνα, η Ινδία, αλλά προσφατά και η Ρωσία, με τρόπο επιθετικό, έχουν εισβάλλει σε εισαγωγικά στην Ευρώπη Οπότε και εμείς θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να δούμε πώς θα αλλάξουμε στρατηγική. Και έτσι να είμαστε αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε προς όφελο της Ευρώπης αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος, η Ευρώπη γυράσκει και όσο αφορά την επιστημονική κοινότητα. Να, κοιτάξτε, το, η ηλικιακή ομάδα 65 συν προβλέπεται να έχει αυξηθεί κατά 20% το 2020 ή μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει το εξή. Θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και να βρούμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς. Να αντικαταστήσουμε πλευράς επαγγελματική και διανοητικής αυτόν τον κόσμο και να μπορέσουμε να βρούμε τους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση που υπάρχει, αλλά επίσης βράχει πρόθεσμα να εξασφαλίσουμε κάποιες δυνατότητες που υπάρχουν για να υπάρχει ανάπτυξη και αντιδραστικότητα στην Ευρώπη. Μια εύκολη λύση είναι το να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τον επαγγελματικό βίο των γυναικών που έχουν αποφυτίσει από πανεπιστήμιο και διαπιστώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι έχουμε 3% περισσότερες αποφύτους πανεπιστήμιων από ότι άντρες. Αλλά λόγω των στερεοτύπων, λόγω των ε, ε, παραδόσεων δεν εκμεταλλευόμαστε αυτές τις δυνατότητες. Το Μακένζι ή ο Μακένζι αναλύει αυτά τα στοιχεία. Είναι Μια επταετία και οπότε θα είπαμε ότι αν μπορέσουμε να καλύψουμε την ε, παραγωγή το 50% αυτών των αποφύτων γυναικών θα έχουν καλύψει το κενό που υπάρχει κατά 3 εκατομμύρια θα το έχουν γεφυρώσει. Και τα είπε η Επίτροπος Κρούς. Μας λείπουν 7.000 ε, καθηγητές πληροφορικής. Έχουμε αυτό το μοντέλο Μακένζι λοιπόν, σύμφωνα με το οποίο 3.035 είναι αυτό το κενό. Οπότε θα φτάσουμε στα 21 εκατομμύρια απασχολήσεις αν συνεχίσουμε και αν ε, κινητοποιήσουμε μόνο τις μισές γυναίκες. Θα έχουμε κενό 3 εκατομμύριων, οπότε τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα καλύψουμε με διάφορα μέτρα. Αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να μας απασχολεί του από τώρα, από σήμερα. Τώρα, για ρίξτε μια ματιά στο τι γίνεται όσον αφορά τις γυναίκες επιχειρηματίες. Υπάρχει ισορροπία στην Ευρώπη μεταξύ εφευρετών, κυρίως στις εφαρμοσμένες επιστήμες, σε σχέση με τις είπα ή την Αφρική. Αν όμως δούμε πιο λεπτομερώς τι δυνατότητες ε, έρευνας υπάρχουν στην Ευρώπη, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε σήμερα 46% των, κατόχων δακτορικών που είναι γυναίκες. Εάν δε, δούμε τι γίνεται όσον αφορά την έρευνα, βλέπουμε ότι μεγαλώνει το χάσμα πάνω από 30% των γυναικών που 30% των, των ερευνητών. Όσον αφορά τώρα τις ανώτερες πανεπιστημιακές θέσεις, οι γυναίκες εκεί είναι το 19,8%, άρα ακόμα λιγότερες, κάτω από το 20%. 15% σαν επικεφαλής διαφόρων ε, ιδρυμάτων, 10% επίσης διευθυντές των πανεπιστημίων, μόνο, στον πρώτο βέβαια πανεπιστήμια, ο ρόλος μου. Δεν είναι να σας πω το πώς θα εξασφαλίσουμε θέσεις για τις γυναίκες. Αλλά θα πρέπει να μας προσφέρουν σοβαρά αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις διανοητικές, πνευματικές ικανότητες, τις ιδέες της Ευρώπης. Και οι ίδια. Είμαι γυναίκα λοιπόν αυτές που, τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες. Να δοθεί ο χώρος, οι δυνατότητες, τα κίνητρα στις γυναίκες να λάβουν πιο πολλές πρωτοβουλίες, ε, πιο ηγετικές θέσεις και έτσι να βοηθηθεί η ανταγωνιστικότητα. Είμαι Βουλγαρά και μπορείτε να δείτε σε αυτά τα στοιχεία ότι η Βουλγαρία υστερεί όσον αφορά την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Δεν επισέρχομαι στις λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Την τελευταία τριετία το μη κυβερνητικέ οργανώσεις, το κράτος, ε, διάφοροι φορείς ακολουθήσαμε μια στρατηγική, ούτω ώστε να έχουμε μια καινούργια προσέγγιση, ένα καινούργιο σύστημα. Να μπορούμε να έχουμε περισσότερη καινοτομία στο μέλλον και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Να είμαστε πρακτικοί στην αντιμετώπιση μας. Ένας από τους τομείς ήταν ε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των πανεπιστημίων. για υψηλή τεχνολογία είπαμε να στηρίξουμε αυτούς που μπαίνουν στην αγορά για, για πρώτη φορά με ειδικά προγράμματα ένα δίκτυο υποστήριξης για τους νέους επαγγελματίες. Αλλά βέβαια προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε αυτή την πολιτική και τα επιστημονικά προγράμματα. Τώρα μπορείτε να δείτε τώρα τι γίνεται με την εκπροσώπηση των γυναικών στην έρευνα στη Βουλγαρία. Τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι υπάρχει γενικά στην Ευρώπη σε μέσο όρο. Ίσως είναι λίγο καλύτερη η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα. Αν δείτε όμως παρακάτω, διαχείριση, διοίκηση ε, ιδρυμάτων επιστημονικών, βλέπουμε ότι είμαστε και εκεί και σε εμά κάτω από το 20%. Κάπως θα πρέπει να ελκύσουμε τις ε, κοπέλες να επιλέξουν ε, τις θετικές επιστήμες. αλλά πιο συγκεκριμένα να επιλέξουν την έρευνα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Έχουμε ε, ένα ίδρυμα όπου έχουμε κάποια σφαιρικά, ολιστικά τα λέμε προγράμματα και εκεί πέρα Ελκύουμε τις νέες επιστήμονες, δίνουν διαλέξεις, μιλούν ενώπιον ακροατηρίων 200-300 ερευνητών και έτσι με αυτόν τον συγκεκριμένο πραγματικό τρόπο προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Έχουν και προγράμματα εκπαιδευτικά. Και συνοδεύουμε τις προσπάθειες από το γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο μέχρι να γίνουν ερευνητές αυτά τα πρόσωπα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το θέμα μας απασχολεί σήμερα, δηλαδή πρώτα πρώτα αυτό που θέλουμε είναι να φτιάξουμε ένα δίκτυο για νέες ε, επιστήμονες οι οποίες να, έχουν ελκυστεί στις ειδικές επιστήμες να προβάλλουμε αυτό το δίκτυο αλλά το σημαντικό είναι να, να, να τις ελκύσουμε σε αυτό το δίκτυο. Ε, επίσης να έχουμε μια υποδομή σε σχέση με τον έφος για τις ΜΜΕ, να υπάρχει τέτοια υποστήριξη για διάφορα τέτοια προϊόντα. Τελικά να πετύχουμε περισσότερη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Μετά από τις τόσο παραγωγικές παρουσιάσεις, να περάσουμε τώρα στη συζήτησή μας, ε, να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Ξεκινούμε από τον κύριο Κλάμπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς ε, μέλη του πάνελ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι τονίσατε τα πιο σημαντικά στοιχεία των ε, συζητήσεων τους τελευταίους μήνες. Το θέμα της απλοποίησης, σχέσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την έρευνα είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και στα οποία συμφωνήσαμε προς τα που θέλουμε να οδεύσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία και την Επιτροπή μας που κατάφερε να συνθέσει με σωστό τρόπο το πάνελ. Κάτι που με ενδιαφέρει επίσης. Μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και για το... την εικόνα που θέλουμε να διέπει αυτόν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Πού θέλουμε να καταλήξουμε. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λένε ότι θέλουμε πολυμορφία 28 μικροί χώροι έρευνας όμως να, θα πρέπει να ενοποιηθούν και να δημιουργηθεί ένας χώρος, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί και η ε, δικαιοδοσία των κρατών μελών. Υπάρχουν και γεωγραφικές ε, διάφορες. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την έρευνα σε περιφέρειες όπου υπάρχει ε, υστέρηση. Θα πρέπει να έχουμε και αυτή την σκάλα, την κλίμακα, αν θέλετε, προς την αριστεία, για να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή, να γίνει εκεί πιο ενδιαφέρουσα η Αυτό λοιπόν θα αποτρέψει και την διαρροή εγκεφάλων. Πού θέλετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία μεταξύ ε, των θεμάτων αυτών. Πού θα πρέπει να θέσουμε τη χρυσή τομή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κούκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές γιατί μας έδωσαν τόσο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μέλλον της έρευνας. Πραγματικά είναι εξαιρετικό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν και κάποιες ερωτήσεις ε, να κάνω. Πώς θέλετε λοιπόν να ανοίξετε αυτές τις κλειστές λέσχες ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία σχετικά. Ξέρουμε όμως ότι στην πράξη τα πράγματα κινούνται διαφορετικά. Καλό θα ήταν να μην τα βλέπουμε όλα αυτά μόνο σε διαφάνειες, αλλά να δούμε και πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά στην πράξη, πώς λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δεύτερη ερώτηση προς τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Ποια είναι η άποψή σας. Ποιες θα είναι οι τεχνολογίες στην Ευρώπη οι οποίες θα είναι οι πιο ανταγωνιστικές. Άλλη μια ερώτηση. Σε ποιους τομείς. Συνολικά. Είναι πιο θετικές οι τάσεις που διακρίνονται από τη δική σας οπτική γωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. πολύ σημαντικές και οι τρεις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση στον ε, καθηγητή Σαλέμα, ο οποίος ήταν σαφέστατος και αποτελεσματικός. Μας είπατε ότι κάποιες τεχνολογίες, εδώ είμαι κύριε Σαλήμα, ε, προέκυψαν από την Ευρώπη και χάρη στη χρήση κοινών προτύπων και ούτε καθεξής και μας έδωσαν ε, στη συνέχεια και κάποιες βιομηχανικές διαδικασίες. Ε, εκεί όμως χάθηκε στη συνέχεια ο ηγετικός ρόλος. Αφού εμείς αποτελέσαμε το έναυσμα, ξεκίνησε η έρευνα, αναφερθήκατε σε διάφορες τέτοιες τεχνολογίες. Και μετά, αναφερόμενο σε κάποιες νέες εφαρμογές, ε, μας είπατε ότι ίσως και εκεί θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε και θα μπορούσαμε να δώσουμε μια νέα όθηση και να κατακτήσουμε και άλλες τεχνολογίες ε, λιγότερο ενεργοβόρες και να μπορέσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστικότητα εχμής σε αυτούς τους τομείς τι χρειάζεται προκειμένου να γίνει αυτό το πέρασμα. Έγιναν ε, οι ανακαλύψεις, έχουμε εντοπίσει σε ποιους τομείς ε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να, ε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε από εκεί και πέρα την κατάλληλη έρευνα και πώς θα το κάνουμε. Ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένως. Αυτές οι ανακαλύψεις της Ευρώπης πώς μπορεί να αποτελέσουν πλαενόκτημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, είτε τη νέα είτε την παλιά και να περάσουν στην παραγωγή ποιο είναι το πέρασμα, ποιο είναι το συγκεκριμένο το οποίο θα πρέπει να γίνει, το οποίο δεν άπτεται πλέον τη έρευνα, είναι άλλα τα μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αν έχετε όμω κάποιε προτάσει επί τη βάση εμπειρία μα, θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο. Ο Βιτόριο Πράντι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, διότι πραγματικά ακούσαμε παρουσιάσεις πολύ πλούσιες, με πολλά στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να αναφερθώ στις προοπτικές της αεροναυτικής. Με τα ηλεκτρικά αεροπλάνα. τα οποία φαντάζομαι ότι θέλουν να, χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιούν ε, καύσιμο ε, κυψέλη, υδρογόνου, επομένως θα έχουμε και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ε, καυσίμου σε σχέση με το παρόν καύσιμο και θα είναι και πολύ μικρότερος ο χώρος ο οποίος καταλαμβάνει στο αεροπλάνο. Πρόκειται λοιπόν για ε, τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά θα είναι ιδιαίτερα παραγωγικές και λυπάμαι που αγνοούσα ότι μέχρι τώρα υπάρχουν ε, πρωτότυπα αεροσκάφη ε, ηλεκτροκίνησης ε, τα οποία ήδη ε, μπορούν να πετάξουν. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική καλή είδηση για τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροναυπηγικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον καθηγητή Σαλέμα, διότι μπορεί να φαίνεται εμένα ότι προκάλεσε μετά τα όσα μας είπε, αλλά η ανωνυμία θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι όποιος καλείται να κρίνει, μου έχει συμβεί και εμένα αυτό, πολλές φορές ε, μένει στα ονόματα και κατά κάποιο τρόπο ε, δεν ε, ε, προσπαθεί να ε, μην σκεφτεί πιο λογικά και δεν αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες. Η πραγματική λοιπόν αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται επί των αποτελεσμάτων όπως είπατε και εσείς και ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται για τα αποτελέσματα και όχι εκ των προτέρων να γίνεται έλεγχος σε οικονομικό επίπεδο για το τι δαπάνες γίνονται και να μην θεωρείται αυτό προτεραιότητα. Όσον αφορά τα όσα μας είπε η κυρία Σάσα Μπεζουχάνοβα, πραγματικά ε, σας ευγνωμονώ ιδιαίτερα. Ίσως εδώ θα πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτή την έρευνα για τις ανθρωπιστικές σπουδέ ε, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν αξιολογήσαμε πλήρως τη συνεισφορά των γυναικών ε, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Και πραγματικά ήταν μεγάλη απώλεια αυτό. Αρκετοί πόροι ε, σπαταλήθηκαν μάταια και νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό και από άλλη σκοπιά. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε μόνο ε, ότι θα πρέπει να είναι τα πάντα επίσης όρις, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τεχνητό. Πρέπει να ξεκινούμε από τη συνειδητοποίηση ότι ο καθένας από εμά μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην πρόοδο. Και επομένως αυτή η ανάγκη να έχουμε προσδοκίες από τους άλλους, ε, προσδοκίες για μια συνεισφορά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη πρόοδος που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε και στη χρήση των πόρων μας εν γέννη. Να περάσουμε λοιπόν σε μια προσδοκία από τους άλλους η οποία θα μας κάνει όλους πιο πλούσιους. Και νομίζω ότι αν κάνουμε αυτό το βήμα θα υπάρχει και αυτή η συνέπεια να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε και πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Κύριε Σαρτόρη, τελειώσαμε με τις παρεμβάσεις. Να δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στους ομιλητές μας για να απαντήσουν. Πέντε λεπτά ο καθής. Ο καθηγητής Μπουργκίνιον καταρχάς. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Υπάρχει μια τελευταία παρέμβαση, ο κύριος Οντή. Ε, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, χρειάστηκε να πουσιάζω στην αίθουσα λόγω κάποιου προσωπικού θέματος και δεν μπόρεσα να ακούσω όλους τους ομιλητές. Διάβασα λίγο τις παρουσιάσεις και θα ήθελα να πω το εξή μόνο. διαρθρωτικό και θεσμικό ζήτημα. Καταρχάς να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας εγώ υπήρξα εισηγητή για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο και εδώ κάναμε μια παρατήρηση για τον πολλαπλασιασμό των μέσων που αφορούν την έρευνα. Εγώ ως Ευρωβουλευτής, ως εκπρόσωπος των πολιτών πρέπει να σας πω ότι ε, πολίτες οι οποίοι δεν είναι φυσικά στο επίπεδό σας ε, των επιτρόπων, των μελών όλων αυτών ε, των επιτροπών Ο τίτλος και μόνο, αν θέλετε, έχει μία υπεροψία ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και οι πολίτες δεν μπορούν να ταυτιστούν ε, Και το διαπιστώσαμε αυτό όταν μιλούν οι ευρωβουλευτές, ε, ακόμα και αυτοί έχουν την εντύπωση ότι ασχολείστε με κάτι πολύ ψηλότερο από αυτό με το οποίο ασχολείστε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ευρωπαϊκή έρευνα. Υπάρχουν δύο ε, υπηρεσίες, υπάρχει εκτελεστική υπηρεσία για την έρευνα, υπάρχει ο δικός σας οργανισμός που ασχολείται με τη δράση, με τον γενικό της διευθυντή και πραγματικά εγώ κάνω έκκληση να σταματήσουν όλοι αυτοί οι τίτλοι, το τάδε κοινό κέντρο έρευνας και το δίνα κοινό κέντρο έρευνας. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προβολή για να γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω πραγματικά, ε, τι να σας πω, αν αλλάξετε το όνομα, διότι ο τίτλος ε, δίνει την... Ε, εντύπωση ότι ασχολείστε με την έρευνα σε υψηλό επίπεδο και μετά διάβασα τι λέει η σελίδα σας στο διαδίκτυο. Φαίνεται να ασχολείστε λίγο πολύ με τα πάντα, μετά μπαίνουμε στη σελίδα και βλέπουμε τι ακριβώς κάνετε. Έκκληση λοιπόν κάνω, πλησιάζουμε σε ευρωεκλογέ και όταν θα προσπαθήσουμε να πλασάρουμε εντό εισαγωγικών την ιδέα ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική έρευνα, όταν θα μα κοιτάξουν οι πολίτε, πραγματικά κανεί δεν θα μπορέσει να του απαντήσει και να μπορέσει να ταυτιστεί με αυτά τα οποία κάνετε. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Ζαμπιέρ Μπουργινιού. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας για το πώς μπορούμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Δύσκολη ερώτηση. από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που λαμβάνουμε για την υποστήριξη τη βασική αυτή έρευνα δεν είναι πολλά. Αυτό όμως είναι ένα μικρό τμήμα. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και να μην έχουμε υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες. Αλλά να σκεφτούμε και το μέλλον. Να γνωρίζουμε προς τα που οδεύουμε. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η υποστήριξη για την έρευνα δεν είναι μόνο ε, οικονομική, χρηματοοικονομική. Το θέμα είναι και να υπάρχουν και θέσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Η οικονομική υποστήριξη της έρευνας τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά και οι σταθερές θέσεις απασχόλησης για τους ερευνητές έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα θέματα αυτά για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας θα πρέπει να τα θεωρήσει κανείς συνολικά. Να μην μιλάμε μόνο για τους πόρους, αλλά και για τον κόσμο, για το πώς διαμορφώνεται το μέλλον των ερευνητών αυτών. Και πολύ φοβάμαι ότι τα τελευταία χρόνια οι τάσεις δεν ήταν ιδιαίτερως θετικές. Υπήρχαν καλοί μαθητές, όπως η Γερμανία, και λιγότερο καλοί μαθητές, όπως άλλες χώρες. Αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της έρευνας στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό συνολικά, όχι μόνο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά συνολικά. Και τώρα... Για τον κύριο Οντή, θα του πω ότι πρώτα-πρώτα δεν ευθυνομαι εγώ για τον τίτλο του Ιδρύματός μας και στη μικρή ιστορική εισαγωγή που έκανα ήταν ε, θαραλέα επιλογή περισσότερων. Και οι βουλευτές είχαν συμμετάσχει. Ήταν ε, οριακή κάλυψη τη συνθήκη για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι τη βασική έρευνα σαν θέμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ερχόμενο σε επαφή με τους ε, επιστήμονες πάρα πολύ λίγοι θα σας πούνε ότι κάποιος που έλαβε μια υποτροφία από το Συμβούλιο δεν έχει αναδειχθεί ε, και πρόκειται για πάρα πολύ βασική και καινοτόμα εισφορά μας. Και οι καλύτεροι επιστήμονες συμμετέχουν στην επιλογή αυτών των υποτρόφων από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο. Τέτοια είναι η συμμετοχή μας στις, στα πάνελ τώρα της επιλογής και 11% προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, πολύ σημαντικό. Και αν δείτε τους εξωτερικούς μας εμπειρογνώμονες, για τις εκθέσει μας έχουμε 89 χώρες που συμμετέχουν Επομένω, Δεν είμαστε σε ένα κλειστό σύστημα πια γίνεται Ευρωπη... μεταξύ Ευρωπαίων. Τώρα όσον αφορά την σαφήνεια. Όχι, δεν τα λέω αυτά επειδή είμαι επικεφαλής του Ιδρύματος, αλλά αν δείτε τι γινόταν στο παρελθόν, τώρα νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο τι γίνεται στον κάθε πυλώνα δράσης. Και επίση για την βασική έρευνα υπάρχει τώρα ξεκάθαρο τοπίο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε επίση την υποτροφία Μαρία ε, πολύ σημαντική για τους νέους Ευρωπαίους ερευνητέ. Επίσης ε, έχουμε τις προσπάθειες που αφορά την κοινωνία ανάλογα για, την, για τον ανταγωνισμό, επομένω νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ε, ο οργανισμός μας. Αντίθετα από το τι ίσχυε προηγουμένως στα πλαίσια του 7ου πρόγραμματος πλαισίου. Τώρα έχουμε πιο συνεκτική προσέγγιση. δε προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτά που κάνει ο Γενικός Διευθυντής, το που κάνει ο Επίτροπος. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμα. Ευρωπαϊκό χώρο έρευνα είναι ο κοινό μα παρονομαστή για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Υπάρχει τεχνολογική πτυχή, οπότε νομίζω ότι όσο πιο σφαιρικά βλέπουμε τα πράγματα, τόσο πιο καλύτερα θα τα πάμε. Όσο μεγάλες και αν είναι κάποιες χώρες, η συνολική προσπάθεια θα πιάσει περισσότερο. Θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Σε αφορά τώρα τις παγκοσμίες τάσεις στην τεχνολογία. Να σα τα πω στα αγγλικά και έτσι θα με καταλάβουν περισσότεροι. That it based on uh, really bottom-up approach. That is the... Η προσεγγίση μας είναι από τη βάση προς την κορυφή. Υπάρχουν προτάσεις και επιλέγουμε τις καλύτερες και έτσι έχουμε αυτές τις επιτροπές επιλογής. Και τα κριτήρια επιλογής είναι πιο σημαντικά από το βιογραφικό ή την προϊστορία του ερευνητή. Να επομένω ότι έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Έτσι δίνουμε κίνητρα τους νέους να υποβάλουν πιο τολμηρές προτάσεις. Η παγκόσμια στάση τώρα στην έρευνα. Έχουν αγγίψει πολλά με πολλούς τρόπους. Κάτι που ίσως θα πρέπει να τονίσω είναι τα δεδομένα. Αυτό που ονομάζουμε μεγάλα δεδομένα. Πολλές επιστήμες βασίζονται εκεί, οργάνωση πόλεων. Τεράστια ποσότητα δεδομένων και για την κλιματική αλλαγή ισχύει. Πρέπει να συλλέξει κανεί τεράστιε ποσότητες δεδομένων, να τα οργανώσει για να γίνουν χρήσιμα. Οπότε και το Ερευνητικό Συμβούλιο προσπαθεί να εξασφαλίσει το ότι η κατανομή στα 25 πάνελ ε, γίνεται σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις. Τα μέλη δουλεύουν μια τετραετία και όχι παραπάνω και φορά προσπαθούμε ακριβώ να εκμεταλλευτούμε τι αντικαταστάσει για να μπορέσουμε να βάλουμε εκεί κάποιου με νέε δεξιότητε και ικανότητε και τα θέματα που καλύπτουν τα πάνελ να παρακολουθούν τι ε, παγκοσμίε τάσει και εξελίξει. Επομένως πρέπει ο καθένας να προσαρμοστεί, να λάβει υπόψη τις νέες τάσεις. Πολύ, πολύ επικαιρό είναι το θέμα αυτό των μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. με τον Ζανπέρ ε, Bourguignon, ο κύριος Μίλλερ Βάισνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι δεν έχω σχόλια για τον κύριο Ντί. Θα ήθελα ως εκπρόσωπος της βιομηχανίας να πω το εξή. Η δική μας εμπειρία την καταδεικνύει ότι όντως ότι το καλύτερο κριτήριο ανάπτυξης είναι τα άτομα. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια στη Γερμανία, νομίζω 12-15 στον αριθμό, για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να δώσω κίνητρα στον κόσμο, να μεταφερθεί σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, να αναπτυχθεί εκεί πέρα η έρευνα και να γίνει μια αρχή. Εδώ συμφωνώ με τον καθηγητή Μπουργκίνιον σε ό,τι αφορά την σημερινή υποδομή. Το θέμα είναι και το βιωτικό επίπεδο. Και αυτό είναι καθήκον των χωρών να το φροντίσουν για να προσελκύσουν τους ερευνητές τα ερευνητικά κέντρα στα οποία συμμετέχουμε ως μέτοχοι σε διάφορες χώρες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα θέμα και πληρωμή των ερευνητών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό με τις ΕΠΑ. Και οι άκαμπτοι κανόνες ε, στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ε, μισθολογικές ε, συμβάσεις. Συχνά συζητάμε πιο πολύ τέτοια θέματα παρά θέματα τεχνικά. Ξέρω ότι παίρνουν χρόνο αυτά, αλλά πραγματικά θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό το θέμα. Ύστερα, τέθηκε ένα ερώτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς θα πρέπει να ανοίξει αυτή η λέσχη. Να πω από πλευράς της δικής μας ε, ε, επιχειρήσεις ότι έχουμε τουλάχιστον τρία εργαλεία για να συνάπτουμε συνεργασίες με νέες μικρές επιχειρήσεις. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη διάσταση των διαγωνισμών, όπου ανοίγουμε τον κύκλο μας σε νέους παροχούς και προμηθευτές, προκειμένου να γνωρίσουμε και τις ε, ενδεχόμενες μελλοντικέ μας ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε συνεργασία και με νέους φορείς. Αν πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους καλούμε να συμμετάσχουν σε έναν όμιλο, προκειμένου να έχουμε έναν εκπρόσωπο του ομίλου αυτού, για να είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία ανάθεσης των έργων. Έχουμε ακόμα και σχετικά μέσα το Aerofund στην Τουλούζη, με το οποίο υποστηρίζουμε την υποστήριξη αυτή από προμηθευτές, προκειμένου να συνεργάζονται και με άλλους ε, προμηθευτές Ακόμα και αν αυτό σημαίνει καθυστέρηση στη διαδικασία ανάθεσης του έργου, προκειμένου να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Υπάρχει ένα άλλο μέσο για την καινοτομία, την οποία τα γνωρίζει απαραίτητα κανείς ιδιαίτερος. Εκεί έχουμε μια διαδικασία με ανοιχτό τέλος, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Δεν έχουμε ακόμα ε, προμηθευτεί τέτοιου ηλεκτρικού κινητήρε για τα αεροσκάφη. Έχουμε κάνει όμω σχετική έρευνα και έχουμε καταλήξει σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, για πολύ, πολύ μικρέ επιχειρήσει, 10-15 άτομα. Την ερώτηση τη κυρία Μερκή. Έχουμε χάσει την ηγεσία και πώς μπορούμε να την ξανακερδίσουμε. Ας πούμε για παράδειγμα ότι κάποιος παράγει λαμπτήρες. 100 βατ. Απαγορεύονται σήμερα έχουμε τα LED. Αυτό το κόστος λοιπόν παραγωγής των λαμπτήρων είναι πάρα πολύ χαμηλό και έχει μεταβερθεί στην Ασία. Γιατί όμως να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γι' αυτό όμως χρειάζεται η έρευνα γιατί την άλλη φορά θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα παράγουν τα LED. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Αυτό που παρήγε κεριά για παράδειγμα, ήρθε σε δυσάρεστη θέση από αυτού που παράγουν λαμπτήρες. Η οικονομική λοιπόν ηγεσία θα πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα, την εφευρετικότητα των επιστημόνων μας, προκειμένου να μην τρέχουμε των υστέρων όταν η μάχη έχει ήδη χαθεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι η ισχύ μα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόντι για τι πολύ καλέ ε, παρατηρήσει για τα ηλεκτρικά αεροπλάνα. Να πω ότι ασφαλώ ε, ερευνούμε και θέματα για την αποθήκευση ενέργειας, αλλά δεν είχα προετοιμαστεί για τεχνικά ζητήματα, για συζήτηση τεχνικών ζητημάτων αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν από δική μου πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Αλέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να δω αν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες για το πώς μπορούμε να συντονίσουμε την ε, έρευνα των κρατών μελών με την ε, έρευνα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας. Να σας πω ότι η ευρωπαϊκή έρευνα το 2020 είναι μόνο περίπου το 5% των ε, ερευνητικών δαπανών στην Ευρώπη. Πώς μπορεί το 5% να συντονίσει το υπόλοιπο 95%? Δεν είναι εύκολο αυτό το ερώτημα. Σίγουρα όχι. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι ο συντονισμός. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να βοηθήσουν. Το δεύτερο ερώτημα ήταν αυτά τα κλειστά κλαμπ. Γιατί υπάρχουν αυτές οι κλειστές λέσχες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μικρά ιδρύματα είναι καταρχάς φοβισμένοι, φοβούνται τη γραφειοκρατία. Πώς μπορούν να υπολογίσουν τις έμεσες δαπάνες, ε, τι θα γίνει με το ΦΠΑ, τι θα γίνει με τις επιλέξιμες δαπάνες. Για μια μικρή επιχείρηση όλα αυτά αποτελούν εφιάλτη. Και φυσικά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ακόμα και η προετοιμασία μιας πρότασης στοιχίζει. Και δεν στοιχίζει λίγα χρήματα στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό. Ένα 20% ε, δαπάνες πρέπει να προβλεφθούν για να υποβάλει κάποιος πέντε προτάσεις υποβολής, ε, ε, υποβολές σε προτάσεις για προσφορές για να μπορέσει να έχει ελπίδες να κερδίσει ένα διαγωνισμό. Και πώς μπορεί να ανοίξει μια χνηστή λέξη, λέσχη. Ε, ένας τρόπος είναι η απλοποίηση. Και τώρα να σας πω κάποια πράγματα από την εμπειρία μου. Ε, προέρχομαι από μια μικρή, όχι και τόσο ανεπτυγμένη χώρα. Πριν από κάποια χώρα διαπιστώσαμε ότι ε, ότι θα πρέπει να βρούμε μια ατμομηχανή. Την αποκαλώ ατμομηχανή γιατί η ατμομηχανή είναι η μεγάλη επιχείρηση η οποία θα σου δώσει ουσιαστικά το εισιτήριο για να συμμετέχει σε μεγάλες διεθνές, διεθνείς προσφορές και να μπορέσει να έχει σε σύμπρεξη και μικρές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η μικρή ε, επιχείρηση μάθει πώς να ελύσεται, ξεπερνάει ένα κατώτατο όριο και μπορεί να προχωρήσει μόνη της. Την πρώτη φορά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά ερευνητικά ιδρύματα. Τρίτον, η αξιολόγηση. Μου δόθηκε εντύπωση ότι έχουμε δύο διαφορετικά προγράμματα. Το ένα είναι η εκ την αξιολόγηση, που είναι η αξιολόγηση της πρότασης, και το άλλο είναι η εκ των υστέρων αξιολόγηση για την παρακολούθηση και να δούμε κατά πόσον ένα πρόγραμμα ε, εκπλήρωσε τους στόχους του. Και εγώ αναφέρθηκα και σε προγράμματα τα οποία εκπληρώνουν τους στόχους τους. Και θα ήθελα να επιμείνω στο εξή: Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ένα πρόγραμμα να πληρεί τις τεχνικές του προδιαγραφές και να μην δαπανά περισσότερο από όσα είχε προβλεφθεί αρχικά. Αν δαπανά κάποιος σε ανθρώπινους πόρους τώρα ή σε οτιδήποτε άλλο, αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία και θα πρέπει να μην μας ενδιαφέρει. Αλλά δυστυχώς ο κανόνας δεν είναι αυτός. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να επιτευθούν οι στόχοι του προγράμματος και επίσης να πληρήσουν τις ε, δαπάνες και να έχουμε ε, μία δήλωση που να έχει ένα προς ένα όλα όσα ξοδέψαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρήσουμε τις προδιαγραφές του προγράμματος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εάν το πρόγραμμα δεν τηρήσει τους στόχους του, τότε σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται και να γίνει οικονομικός έλεγχος. Και τέλος, η πιο δύσκολη, η χειρότερη ερώτηση νομίζω που μου θέσατε είναι πώς να μπορέσει η Ευρώπη να αξιοποιήσει η ίδια τις ανακαλύψεις της. Πώς να ε, πληρώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει από την έρευνα στην αγορά. Πολύ δύσκολη ερώτηση, δεν είμαι εγώ κατάλληλος για να σας απαντήσει, αλλά μια-δυο ιδέες. Καταρχάς, να δώσουμε μάχη για ευρωπαϊκές προδιαγραφές παντού. Αν η Ευρώπη τηρήσει τις δικές της προδιαγραφές, θα τα καταφέρει. Το GSM νομίζω ότι αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα. Όλη η Ευρώπη συγκεντρώθηκε και ενέκρινε το GSM. Μετά είχαμε το DVB, τα βίντεο. Και πάλι η Ευρώπη έκατσε, συνεργάστηκε, αλλά δεν τα κατάφερε ε, σε άλλα στοιχεία. Να σας δώσω και κάτι ακόμα το οποίο αναφέρεται εδώ σήμερα. Η ασφάλεια η ασφάλεια και η ιδιωτική, ε, προστασία της ιδιωτικής ζωής στις επικοινωνίες. Η Ευρώπη ανοίγει το δρόμο, έχει ηγετικό ρόλο και έχει κάποιες ε, ε, συσκευές ασφαλείας κβαντικές, τις οποίες μπορεί κάποιος να τις αγοράσει και να τις εγκαταστήσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι φθηνό, δεν λέω ότι είναι ε, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εν μία νυχτή. Αλλά υπάρχει. Και η Ευρώπη, εάν έχει δικέ τη προδιαγραφέ, τότε σίγουρα θα έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό. Αρχίζουν σιγά σιγά όμω, αν αρχίσουν σιγά σιγά να ε, υπάρχουν διάφορε προδιαγραφέ παντού, θα χαθεί η αγορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα όταν δεν υπάρχει ενιαία αγορά αν υπάρχει ενιαία αγορά και ενιαίος τρόπος έγκρισης προδιαγραφών, νομίζω ότι η ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να ε, έχει ευρωπαϊκά προϊόντα στην αγορά, να μετατραπεί σε ευρωπαϊκά προϊόντα στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαλέμα και τέλος μια τελευταία παρέμβαση και μετά θα μιλήσει κάποιος συνάδελφος. Το λόγο έχει η Σάσα Μπεζουχάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Actually, uh, I think uh, speaking about uh, Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση στην Ευρώπη. Πώς η έρευνα θα γίνει αποτελεσματική. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο επίγουν τα πράγματα Να δούμε. Με τι τρόπο θα το πετύχουμε αυτό. Να το δούμε και θεωρητικά και πρακτικά. Για την νέα περίοδο προγραμματισμού η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή είναι ο πιο δημοκρατικός τρόπος. Έτσι έχουμε την ελευθερία για να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Και έτσι μπορούμε να έχουμε κάποιους, ε, κάποιους τομείς όπου μπορούμε να έχουμε κάποιους κανόνες που να είναι όχι πανευρωπαϊκοί, να έχουν ένα συγκεκριμένο ενιαίο πλαίσιο για την πνευματική διοκτησία, πρώτα-πρώτα. Μιλήσαμε για, τους, για τον μεγάλο όγκο δεδομένων, τις μεγάλες ομάδες τους είπαν δεδομένων. Αυτό αφορά κάθε είδους ε, έρευνα. Οι νέες ιδέες, οι νέοι εφευρέτες, θα πρέπει να καταφύγουν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Σαν Φρανσίσκο για να κατοχυρώσουν αυτό που βρήκαν. Και έτσι, να δούμε πώς θα διορθωθεί αυτή η προσπάθεια κατά τον καλύτερο τρόπο. Ένα άλλο θέμα τώρα. Πώς θα εξασφαλιστούν μηχανισμούς αποτελεσματικούς για την ανταλλαγή των πληροφοριών, για αυτούς που ξεκινούν μια προσπάθεια στον επιχειρηματικό χώρο. Τα κέντρα αριστείας είναι επίσης πάρα πολύ καλός τρόπος, αλλά επίσης για την έρευνα έχουμε σήμερα αυτούς τους αυτούς τους εικονικούς άλλους τρόπους. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι πιο αποτελεσματικέ οι γυναίκες, τα προγράμματα για τις γυναίκες. Έχουμε μία σειρά μελετών, κύριε πρόεδρε γι' αυτό. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας. για τις γυναίκες και την εμπλοκή του στην έρευνα. Θεωρώ ότι σήμερα είναι κάπως μια κλειστή λέσχη η έρευνα και τι αποφάσει δεν τι λαμβάνουν οι γυναίκε. Επομένω, χρειάζεται να δούμε πώ θα μπλοκούν προ γυναίκε, πώ οι γυναίκε θα καταλάβουν, θα, θα μπουν περισσότερο στην υπόθεση των ηγετικών, των διευθυντικών θέσεων. Και να καλυφθούν από κάποια προγράμματα και έτσι να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός που να είναι ελκυστικός και σε αυτό το επίπεδο. Αυτά για το συζήτησή μας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λάγκεν. Σα ευχαριστώ και λυπάμαι που ζήτησα το λόγο τόσο καθυστερημένα. Στην αρχή ήθελα να ακούσω μόνο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αρκετές απαντήσεις, ωστόσο έχω και μία ερώτηση την οποία θα ήθελα να θέσω συμπληρωματικά προς όλους τους ε, καλεσμένους μας. Το θέμα των διαφορετικών ορισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα αποτελεί απόρρια 28 εθνικών συστημάτων. Ο πρόεδρο, η μας και οι συνάδελφοι από άλλε ομάδε. όρισαν τα πράγματα λίγο διαφορετικά είπατε για τον ευρωπαϊκό χώρο ε, έρευνας είναι ο, η οδός προς το Μάστρεχτ. Το Μάστρεχτ είναι η ευρωπαϊκή διάσταση, εναρμόνιση των ε, προδιαγραφών, των ορισμών, των ε, κανονισμών προώθησης. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να ισχύσει γιατί η ισχύς έγκυται στην πολυμορφία, στην ανοιχτή επικοινωνία, στον ανοιχτό διάλογο των διαφορετικών συστημάτων και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πούν τα μέλη του πάνελ πώς εκτιμούν το θέμα αυτό, γιατί δεν συμφωνώ με μια μαζική κεντρική διάσταση, μια, ένα, μια ενιαία διαμόρφωση. Φτάνει πια η ενιαία διαμόρφωση. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει διάλογος, ανταγωνισμός. Όχι να κάνουμε την ίδια έρευνα πολλές φορές, αλλά να μην υπάρχει ένα μοντέλο αλλά Maastricht τύπου ευρώ. Αυτό θα με βρίσκει κάθετα αντίθετο και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη από αυτού. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Λάγκεν. Μία ερώτηση έχουμε. Αν ένας ευρωπαϊκός χώρος ε, έρευνας είναι αυτός ο οποίος μας αρμόζει ή 28 εναρμενισμένα συστήματα. Σύντομες απαντήσεις ο κύριος Μπουργκινών καταρχάς. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα και ξέρετε ότι είμαι μαθηματικός. Χωρίς ορισμούς λοιπόν δεν μπορώ να εργαστώ. Για το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι καταρχάς ότι για τους επιστήμονες είναι ξεκάθαρο. Τα κανονικά όρια, τα πολιτικά όρια ενδεχομένω να μην υπάρχουν. Είμαστε συνηθισμένοι να λειτουργούμε σε διάφορα συστήματα. Αν γράφετε κι εσείς μια έκθεση για κάποιο θέμα, μπορείτε να την καταρτίζετε για διάφορες χώρες και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ποιότητα της εργασίας Και ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες είναι διαφορετική η όρη προώθησης, αλλά αυτό ίσως να δίνει δυνατότητα, να μην παρεμποδίζει τη δυνατότητα μετακίνησης των ερευνητών. Τι χρειαζόμαστε όμως, αυτή είναι η συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι το εξή. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι αρκετά συμβατοί προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του δραστηριότητα σε διάφορες χώρες. Και ξέρετε ότι σε αυτό συγκαταλέγονται και οι κανόνες για τη συνταξιοδότηση, Δεν νομίζω ότι η απάντηση είναι να γίνουν όλα ενιαία και ίδια. Όχι. Αλλά να υπάρχει συμβατότητα και ξέρω ότι σήμερα δεν υπάρχει επαρκή συμβατότητα. Αυτό ενδεχομένω να μπορεί να έλθει από την Ευρώπη. Και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι και το Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί να ορίσει ποιοι είναι οι όροι εκείνοι τους οποίους θα πρέπει να πληρεί κανεί προκειμένου η συμβατότητα αυτή να είναι εφικτή στην πράξη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα και σίγουρα προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε. Όχι, λοιπόν, εξίσωση, καθολική, αλλά συμβατότητα. Για να πετύχουμε τη συμβατότητα αυτή δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. Κύριε. Κύριε Λάγκε, εγώ ως εκπρόσωπος της βιομηχανίας δεν μπορώ να προδιαγράψω του ορισμού για το Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η δική, μου, η δική μας εταιρεία 150.000 εργαζόμενοι, 5.000 ερευνητέ διαδραματίζει ρόλο σημαντικό σε διάφορες χώρες. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά, έχουμε το ίδιο όραμα. Τι χρειαζόμαστε, ε, μία δημιουργικότητα από κάτω προς τα πάνω, γιατί η δύναμη των πολλών είναι πάντα μεγαλύτερη από το μονομένο άτομο. Αλλά σε μια εταιρεία όπως η δική μας χρειαζόμαστε και μια στρατηγική από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχει λοιπόν στρατηγική ατζέντα στις διάφορες χώρες, στην Γερμανία, στην Γαλλία. Ο συνδυασμός λοιπόν των δύο αυτών στοιχείων, θα συμφωνήσω και με τον ε, κύριο Μπουργκινιό, είναι απαραίτητος, αλλά να μην εξισωθούν όλα, να μην μπουν όλα στον ίδιο κουβά. Γιατί αυτό θεωρώ ότι θα παρεμπόδισε τη δημιουργία νέα γνώση. Α, ένα σημείο ακόμα, επιτρέψτε μου. Το θέμα του ελέγχου των εξαγωγών. Μιλώντα για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα, αυτό δεν έχει να κάνει με το στρατιωτικό σκέλο. Κάθε χώρα έχει ένα τέτοιο έλεγχο. Και αν ένα πολιτικό θέμα, ένα θέμα που απαιτείται τη πολιτική διάσταση θέλει να συζητηθεί, θα πρέπει να περάσει από το θεωρητικό έλεγχο. Πρώτα να δούμε κατά πόσον υπάρχει τέτοια ευαισθησία ή όχι για να υπάρχει αυτή η εξαγωγή. Ο κύριος Αλένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, από τη φύση της έχει διεθνή χαρακτήρα η επιστήμη, άρα η πρόοδος απαιτεί ελευθερία για την επιστήμη. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε ομοιομορφία. Τουλάχιστον δική μου γνώμη αυτή είναι, δεν γίνεται. Βεβαίω πολλά μπορεί να γίνει, να έχουμε κάποιε διαδικασίε οι οποίε να προσωμιάζουν να είναι συμβατέ. Και φυσικά έχουμε μάθει πάρα πολλά. υποβάλλοντας προτάσεις... και στη διαδικασία μαθαίνουμε, μαθαίνουμε πολλά. Μαθαίνουμε τι πάει να πει. Ε, συντονισμός αυτό είναι. Μπες δεν θα διαφωνήσουμε με του συναδέλφου που έλαβαν τον λόγο προηγουμένω βεβαίω και χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε κάποια κοινά πρότυπα και του μηχανισμού να είναι συμβατά. Και έτσι έχουμε το πλεονέκτημα του συντονισμού. Και δεν άγγιμα σε σχέση με αυτό που εσείς ρωτήσατε, ναι, είμαι υπέρ τη ποικιλία των προγραμμάτων και έτσι να έχουμε ένα πλαίσιο, μια ατζέντα για την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει πάντοτε να αφήνουμε χώρο για την δημιουργικότητα. Για το να υπάρχει περιθώριο επιλογής θεμάτων που να επιδέχονται συνεργασία πανευρωπαϊκή. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός. Α, και εγώ που είμαι από νέο κράτος μέλος. Η εντύπωσή μου είναι θα από μια δεκαετία θα έχουμε πλέον έκτημα. Α, θα έχουμε αντιλήσει πλέον έκτημα για όσα τώρα δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί. Αυτό θα βελτιώσει πολύ τα πράγματα, να βρούμε δηλαδή κάποια τέτοια πρότυπα. Να μπορέσουμε έτσι να επισημάνουμε ακριβώς ποιοι είναι οι συντελεστές να ελκύσουμε νέους και γυναίκες αυτό ακριβώς για το οποίο μίλησα σήμερα. Καλώς λέει πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε λοιπόν σήμερα το πρωί. Συνεχίζουμε στις 3. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας, τον κύριο Μπουργκινιόν, τον κύριο Μίλερ Βιέσνερ, τον κύριο Σαλέμα και την κυρία Μπεζουχάνοβα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Καλό μεσημέρι.